Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίου για την αξιολόγηση και το συντονισμό των θεμάτων ασφαλείας και το άρθρο 70 και την κατάσταση στη Europol και στη Eurojust. Πρέπει να σας πω ότι τα... έχουμε μία κατάσταση ανάλογα με το άρθρο 70-71 και 85 και 86 διότι το άρθρο 70 λέγεται, λέγει ότι ε, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να αξιολογήσουν αυτές τις ε, πολιτικές ενώ τα άρθρα 85 και 88 λέει ε, ότι είναι προαιρετικό και υπάρχει μία διάκριση μεταξύ των δύο. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα συμμετάσχουν εις την αξιολόγηση αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο δεν μπορούμε εμείς να επιλύσουμε. Το τελευταίο θέμα, η τελευταία ερώτηση αναφέρεται στα συμπεράσματα των διεθνών ε, ε, συμφωνιών ε, για τα άρθρα 24 και 38 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν χρειάζεται ε, συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά αυτό θα αλλάξει άπαξη ισχύ στη συνθήκη της Λισαβόνας και η απόφαση απλά είναι ότι αν οι συμφωνίες έχουν συναυθεί πριν την ισχύ της συνθήκης δεν χρειάζεται η συνένεση του Κοινοβουλίου εάν ισχύσουν όμως μετά από την έναρξη της ισχύω θα χρειαστεί η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με συγχωρείτε η σύναψη μια συμφωνίας καλύπτει και την κύρωση. Δηλαδή θεωρούνται ότι έχουν ε, ολοκληρωθεί, συναφθεί, ε, άπαξ και έχουν κυρωθεί. Ε, βέβαια η, κατάληξη είναι η κύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά δεν είναι το ίδιο και ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια. Εδώ όταν μιλάμε για conclusion μιλάμε για υιοθέτηση της ε, συμφωνίας για εσωτερική νομοθεσία. Άπαξε συναφεί συναφή μια συμφωνία αλλάζει κατάσταση αναλόγως του καθεστώτος υπό το οποίο τελεί παλαιό ή καινούριο καθεστώς. Όσον αφορά τις διατάξεις της συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την σύναψη. Πρέπει πρώτα να συναφθεί η συμφωνία και μετά απορρέουν όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κάλυψα και τα 12 ερωτήματα που τέθηκαν σήμερα το πρωί στην νομική υπηρεσία και όπως σας είπα τις ε, απάντησα εντάχει και αν μπορώ να βοηθήσω μπορώ να σας πω και κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ήδη τρεις αιτήσει λόγου και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους διότι ήδη στο πρώτο θέμα ήδη έχουμε καθυστερήσει παρακαλώ λοιπόν τους παρεμβαίνοντες να είναι σύντομοι και να μην υπερβούν τα δύο λεπτά. Στη συνέχεια, μετά το γύρο των ερωτήσεων, θα επανέλθουμε στην νομική υπηρεσία και θα παρακαλέσω και το Συμβόλιο, Συμβούλιο να ε, εξετάσει ε, τι ήταν ε, η κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής που σήμερα έχουμε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση και ευχαριστώ για τις προκαταρτικές εξηγήσεις. Εγώ ε, αναφέρομαι στην απελευθέρωση των θεωρήσεων προς τις τρίτες χώρες διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει μεγάλες ανησυχίες ε, σχετικά με αυτή την έκθεση και την έκβασή της και άκουσα ότι ε, εάν το Συμβούλιο υιοθετήσει την έκθεση αυτή την τελευταία μέρα του Νοεμβρίου είναι αρκετό και χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα για να ισχύσει αυτή η έκθεση. Αναφέρομαι στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο και στην ΦΥΡΟΜ η οποία πρόκειται να ξεκινήσουν τη συνεργασία ε, την 1η Ιανουαρίου και ε, θα ψηφιστεί η απόφαση 12 Νοεμβρίου ε, θα μπορέσει λοιπόν να ισχύσει ο κανονισμός την 1η Δεκεμβρίου. Θα ήθελα να μου απαντήσει το Συμβούλιο αν οι πληροφορίες αυτές οι οποίες μου έχουν δοθεί είναι σωστές, αν ε, όντως έτσι έχει κατάσταση, εάν ε, το Συμβούλιο θα μπορέσει να ψηφίσει το θέμα αυτό την τελευταία μέρα του Νοεμβρίου αν δεν ψηφιστεί τότε αν επαρκεί για τις τρεις χώρες να μπορέσουν ε, να έχουν απαλλαγή θεωρήσεων από τις 1 η Ιανουαρίου διότι όπως ξέρετε αυτό επηρεάζει πολλοί τους πολίτες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ αυτής της καταργήσεως των θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Η Σάρα Λάτφορντ είναι η επόμενη. Αναρωτιέμαι αν η νομική επιτροπή, η νομική υπηρεσία μπορεί να μου πει αν μπορεί να υπάρξει νομική συνεργασία εφόσον αν τώρα 1η Δεκεμβρίου ισχύσει η συνθήκη, ε, αν υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών ή του Συμβουλίου να ενεργήσουν κατά τρόπον ώστε να μην υπονομεύσουν ε, τις διατάξεις της συνθήκης. Δηλαδή ε, παραδείγματος χάρη ένας τομέας ε, όπου καλό θα ήταν ε, να οργανώσουν μία ημερομηνία συνεδριάσεως πιο πριν αλλά υπό άλλους όρους μπορεί να θεωρηθεί ότι προσπαθούν να τορπιλήσουν το όλο θέμα της συνθήκης. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση ή απλώς πολιτική καλή πίστη για να προχωρήσει το θέμα. Ε, υπάρχει νομική καλή πίστη η οποία να απαιτείται από το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Είμαι πεπισμένη ότι το Συμβούλιο θα ενθουσιαστεί να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να απαντήσει το Συμβούλιο. Ε, ο κ. Μπουσουτήλ, θέλω να καλωσορίσω την επερχόμενη συνθήκη της Λισαβόνας και ευχαριστώ ε, τον κύριο Κλάους που υπέγραψε και χθε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπράτλι για τις ε, λεπτομερείς εξηγήσεις του. Ε, χαίρομαι που έχουμε κάποιον σαν κι αυτόν για να μας δώσει την νομική του συμβουλή. Να ρωτήσω κάτι. Θα θέλαμε όλα αυτά να τα λάβουμε γραπτός, Πρόεδρε. Γιατί δεν τα κατάλαβα όλα. Δεν κατάλαβα όλες τις απαντήσεις, όλες τις ερωτήσεις και φαντάζομαι ότι ισχύει για πολλού συναδέλφους το ίδιο σε σχέση με τα υπάρχοντα θέματα, τους υπάρχοντες φακέλους. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Θα πρέπει να βρούμε ένα πρακτικό τρόπο για τους βουλευτές προκειμένου να καταλαβαίνουν πάρα αυτά. Ποιο τμήμα της ημερήσιας διάταξης άλλαξε, η νομική, άλλαξε και μάλιστα άλλαξε η νομική του βάση και πώς άλλαξε. Είναι ένα ερώτημα πρακτικής φύσης. Ε, κάνω και έκκληση στην γραμματεία να μας βοηθήσετε, να μας δώσετε μια κατεύθυνση, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως για του ισχύοντες φακέλου, για τους φακέλου που τρέχουν. Αλλιώς πραγματικά θα μπερδευτούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν πολλοί μαζί σας, αν όχι όλοι. Ε, ενημερώθηκα ήδη από τη γραμματεία ότι ένας κατάλογος θα κυκλοφορήσει αύριο και είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Μπράντλι θα μας δώσει και γραπτός ε, τις απαντήσεις του. Ναι, γνέφηκε καταφατικά. Βάλτε για κάποιους υποτίτλους σας παρακαλώ για εκείνους που δεν είναι πολύ επαΐοντες στα νομικά για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Ο κύριος Λαμπρινίδης. Ένα ερώτημα για το 4, για τα εθνικά κοινοβούλια και την αρχή της επικουρικότητας. Η νέα συνθήκη δίνει 8 εβδομάδε από την ε, αρχή τη νομοθετική διαδικασία. Όχι από το τέλο τη, όχι από την υιοθέτηση τη νομοθετική πράξη, από την αρχή τη διαδικασία. Τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν 8 εβδομάδε για να σχολιάσουν λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, το μόνο ερώτημα στον κατάλογο των ερωτήσεών μα είναι αυτό για το οποίο η νομική υπηρεσία μοιάζει να υπονοεί ότι αν κάτι έχει ολοκληρωθεί πριν από τη θέση ισχύ τη νέα συνθήκη, παρόλα αυτά οι νέοι κανόνες θα ισχύουν. Και αυτό τι σημαίνει. Ότι αν μια νομοθετική διαδικασία έχει ξεκινήσει, ας πούμε, 10 εβδομάδε. εδώ και 10 εβδομάδες, έτσι. Αν η νέα συνθήκη τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, λέει η νομική υπηρεσία τι, ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν το δικαίωμα τότε να σχολιάσουν αυτή τη διαδικασία παρότι έχουν, έχει περατωθεί η προθεσμία των 8 εβδομάδων. Γιατί μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε εμείς και φυσικά να το καταλάβουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, δύσκολα αυτά τα θέματα για όλους μας. Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι. Πριν δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μπράτλι, θα ήθελα να κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις. Για το τελευταίο θέμα. Όλες οι εκκρεμεί διαδικασίες, εκείνες δηλαδή που, δεν, που έχουν ξεκινήσει και που δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα ξαναρχίσουν. Έτσι. Και, αυτή... και έτσι θα συνεχιστούν αυτά τα πράγματα. Αυτή η διάταξη θα ισχύει. Τώρα, το ερώτημά μου είναι, ε, επειδή ασχολούμαι με το θέμα PNR, με ενδιαφέρουν οι διαδικασίε που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η συμφωνία με τι ΗΠΑ ισχύει προσωρινά, δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, μπορεί να μην είναι τμήμα της διαδικασίας αυτό, αυτό καθ' αυτό, αλλά αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί. Και επομένω θα πρέπει να τύχει επαναδιαπραγμάτευση ή να την να ξεχάσουμε εντελώ. Λοιπόν, αυτέ είναι οι ερωτήσει μου και θα ήθελα μετά, αφού απαντήσετε, να σχολιάσει το Συμβούλιο. Πρόεδρε τα συμπληρωματικά ε, ερωτήματα είναι πολύ ειδική φύσεω. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να σα απαντήσω γραπτό σε αυτά, αν δεν έχετε αντίρρηση. Νομίζω είναι ο καλύτερο τρόπο για να ενημερώσω την Επιτροπή. Ε, το ερώτημα του κυρίου Λαμπρινίδη συζητείται εδώ και καιρό και επομένω. Δεν έχουν αποφασίσει οι νομικές υπηρεσίες των ε, οργάνων για τις προσωρινές, ε, την προσωρινή ισχύ των συμφωνιών θα πρέπει να το κοιτάξω πάντως. Ε, εγώ λοιπόν, επειδή για προσωπικούς λόγους ήρθα σήμερα το πρωί, ε, είχα πολύ λίγο χρόνο για να εξετάσω αυτά τα θέματα. Δώστε μου λίγο χρόνο για να τα κοιτάξω και να σας απαντήσω γραπτός. Πολύ ωραία. Βλέπω ότι η διαδικασία επιταχύνεται. Θα θέλαμε να μας δώσετε τουλάχιστον γραπτός τις απαντήσεις που μας ε, παρουσιάσατε προφορικά πριν από λίγο. Ε, φαντάζομαι τα έχετε κιόλα σε χάρτου. Σας παρακαλώ λοιπόν μοιράστε τα αντίτυπα αυτά και, και για τις επιπρόσθετες ερωτήσεις θα ήθελα να μας απαντήσετε μέχρι αύριο, αν γίνεται. Γίνεται? Έχω την αίσθηση ότι δεν με ακούτε. Δεν ακούγεται η φωνή μου πάλι. Μ' ακούτε? Δεν ακούγομαι, λέει η Πρόεδρος προς τους τεχνικούς. Να απαντήσω εγώ, λέει ο κ. Μπράντλι. Φυσικά θα συνεργαστούμε. Όλοι οι πάλι συνεργαζόμαστε. Πρόεδρε, και κόβεται ο κύριος Μπράντλι. Δεν θα σας εγγύθω ότι θα είμαι έτοιμο ε, με τις απαντήσεις ε, αύριο. Αλλά θα... Επειδή έχω και άλλες ερωτήσεις να απαντήσω στην Επιτροπή σας μέχρι αύριο, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό να μου ζητάτε μέχρι αύριο να απαντήσω σε αυτές τις επιπρόσθετες ερωτήσεις. Ο ήχος μειώνεται, η ένταση του ήχου μειώνεται. Μ' ακούτε τελικά ή δεν μ' ακούτε. Βάλτε όσοι έχετε ακουστικά. Τέλο πάντων, δώστε μου το συντομότερο δυνατόν τι απαντήσει. Ξέρω ότι θα, είμαστε, θα πάντα στο πλευρό μας, ε, έτοιμος να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Τώρα, δίνω το λόγο στο Συμβούλιο για να μας πει πώς βλέπει την επόμενη περίοδο, τις επόμενες εβδομάδε και μήνες. Οι διαδικασίες οι οποίες ε, τρέχουν και για τις οποίες υπάρχει προθεσμία πολύ κοντά στην ημερομηνία που προβλέπεται σε για την έναξη συνθήκης της Λισαβόνας τώρα Συμβούλιο είσαστε σε θέση, γιατί δεν είσαστε την περασμένη εβδομάδα, να δώσετε στο Κοινοβούλιο περισσότερο χρόνο και να ξεκινήσει η διαδικασία εκ νέου υπό τη νέα συμφωνία. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. Όπως και εσείς, η Σουηδική Προεδρία καλωσορίζει την υπογραφή και πιθανότατα θα ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου η συνθήκη. και τότε από την 1η Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτήν. Τώρα στην πράξη αυτό σημαίνει ότι σε ό,τι φορά το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων και άλλα ζητήματα που εκκρεμούν η απόφαση προβλέπεται για τις 13 Νοεμβρίου και θα θέλαμε οι αποφάσεις αυτές να ληφθούν την, 13, την 30 συγγνώμη, Νοεμβρίου. για να μην χαθούν ε, κάποιες ευκαιρίες. Η Προεδρία λοιπόν θα ήθελε να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει το συντομό των δυνατών ώστε να μπορέσουν να εγκριθούν οι αποφάσεις πριν από σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνας. Όταν όμως πρόκειται για ζητήματα των οποίων προθεσμίες έχουν οριστεί για τον Δεκέμβριο τότε θα αναγκαστικά θα βρεθούμε στο πλαίσιο της Θήκης Λισαβόνας και ελπίζουμε οι εργασίες που θα έχουν γίνει μέχρι τότε και που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό στο Συμβούλιο θα ληφθούν υπόψη όταν οι νέες προτάσεις υποβληθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νέα συνθήκη. Θέλουμε να κάνουμε λοιπόν διάκριση ανάμεσα σε κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε αποφάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα συνθήκες και άλλες ε, να ληφθούν σύμφωνα με την Λισαβόνα, περιμένοντας τις ε, προτάσεις. Η Κομισιόν σε αυτές περιπτώσεις αλλά και σε άλλες όπως αναφέρθηκε θεωρεί ότι αυτό είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Οι προθεσμίες του Συμβουλίου δεν πρόκειται να τροποποιηθούν αυτές συνεχίζουν να ισχύουν και δεν προβλέπεται να αλλάξουν οι ημερομηνίε συνεδριάσεως του Συμβουλίου. Προς τον παρόν αυτά έχω να πω. Αυτό σημαίνει πως σε ορισμένους φακέλους θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας σύμφωνα με τη νέα συνθήκη ενώ οι άλλες περιπτώσεις θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Πρόεδρος, διακρίνεται ανάμεσα στις διαδικασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν πριν από την 1η Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία. Και διαδικασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά. εδώ δεν έχουμε και πολλές ε, επιλογές. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι οι διαδικασίες επί των οποίων το Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμα πάρει θέση και είναι μάλλον απίθανο να λάβουμε θέση μέχρι τα τέλη του μήνα όπως το ζήτημα της Europol αλλά και άλλες. Αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα και θα ήταν ζήτημα ευγένειας από πλευρά ε, Συμβουλίου να αναγνωρίσει πως ε, θα πρέπει από τώρα να ενεργούμε στο πλαίσιο, ε, στο πνεύμα μάλλον της Δίκης Λισαβόνας και Εάν ε, το Συμβούλιο επιθυμεί να ξεκινήσουν αυτές οι διακές που δεν έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη Λισαβόνας, ε, μπορούσε να μας το αναφέρετε αυτό. Έκανε διάκριση σε, για τους φακέλους ε, για τους οποίους προβλέπεται ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, τότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην υιοθέτησή τους. Άλλο το παράδειγμα όμως των δικονομικών θεμάτων που εκκρεμούν, τότε αυτά θα πρέπει να προωθούν μέσω της συνήκης της ε, Λισαβόνας. Αυτή είναι μια διάκριση που θα προσπάθησα να σας κάνω. Ελπίζω τώρα να είμαι σαφέστερη. Λοιπόν, να Βλέπω ότι ορισμένοι έχουν σηκώσει το χέρι τους και έχουμε διαδικασίες χωρίς χρόνο να απαντήσουμε. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να βιαστούμε τόσο πολύ για ορισμένους φακέλους. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να υιοθετηθούν ταχαίως, αλλά για άλλους δεν βλέπω γιατί υπάρχει και βία να υιοθετηθούν πριν την 1η Δεκεμβρίου, εκτός και αν το Συμβούλιο θέλει να αποκλείσει το Κοινοβούλιο εσκεμένος είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να γνωρίζω. Δηλαδή, ορισμένες διαδικασίες γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν 1η ε, Δεκεμβρίου. Ο κύριος Άλμπρεχτ και η Σάρα Λάτρο ζητούν το λόγο και για μένα η κατάσταση είναι κάπως συγκεχημένη διότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε αυτή τη συζήτηση ε, εάν δηλαδή είναι όντως απαραίτητο να ληφθεί αυτή η απόφαση για την Europol πριν από το τέλος του χρόνου και δεν ακούσαμε κάποιο επιχείρημα υπέρ και τώρα μας λένε 1η ε, Δεκεμβρίου, δηλαδή ε, πέντε ημέρες ε, μετά την υιοθέτηση της αποφάσεως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακόμη δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 1η Δεκεμβρίου και νομίζω ότι όντως μας συμπεριφέρονται διότι το Συμβούλιο δεν ε, προσβλέπει καθόλου στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μήπως το Συμβούλιο μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξει αναβολή και θα υπάρξει μία ρύθμιση και θα υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες θα υιοθετηθούν μόνο εφόσον είναι απαραίτητο και η διαδικασία θα μπορέσει να ανακοινηθεί πάλι υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Η Σάρα εάν κατάλαβα καλά. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν περιοχές ασάφειας, αλλά το Συμβούλιο εδώ μας παραπέμπει σε περιπτώσεις όπου η γνωμοδότησή μας θα υπερβεί το τρίμηνο της προθεσμίας που έχει καθορίσει το Συμβούλιο, άρα ε, θα μπορούσε θεωρητικά ε, το Συμβούλιο να υιοθετήσει ένα μέτρο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ακόμη και αν δεν έχει γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν το Συμβούλιο προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο ή θα κινηθεί σε ένα πνεύμα τίμιας συνεργασίας πέραν των νομικών υποχρεώσεων και θα πει ότι αναγνωρίζουμε ότι πολιτικά αν όχι νομικά δεν θα ήταν σωστό να ε, αποδεχθούμε κάτι το οποίο νομικά θα μπορούσαμε αλλά το νεοεκλεγέν κοινοβούλιο που έχασε τρεις μήνες και δεν είχε επαρκή χρόνο να οργανωθεί για να εκδώσει την απόφασή του εντός ε, τριμηνίας θα αγνοηθεί. Δηλαδή βάσει τεχνικών επιχειρημάτων να περιοριστεί κανείς στο τρίμηνο. Το σύμβολο μπορεί να μας πει αν όντως η κατάσταση έτσι έχει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, κύριος Μπουσουτήλ ίσως έχουμε υπάρξει κάπως άδικοι προς το Συμβούλιο και αν είναι ευγενεί προς εμάς θα έπρεπε και εμείς να τα αποδώσουμε. Άρα ας εξετάσουμε περίπτωση κατά περίπτωση που υπάρχουν φάκελοι οι οποίοι εκρεμούν ακόμη και κατά περίπτωση να εξετάσουμε τι μπορεί να γίνει. Προτείνω λοιπόν στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών, δηλαδή αν είναι δυνατόν αύριο, να έχουμε έναν σαφή κατάλογο των φακέλων όπου πλησιάζει ε, ε, το κλείσιμό τους, διότι ε, διαφορετικά δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν ούτως ή άλλως. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στους φακέλους όπου εύλογα Πιστεύουμε ότι μπορούν να ολοκληρωθούν αυτό το μήνα και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε κατά περίπτωση και μόνο κατά περίπτωση ακόμη και αν α, επαναλαμβάνουμε μπορεί κανείς να πει ότι θα αξιολογήσει πολιτικά τις περιπτώσεις. Ε, μην πούμε λοιπόν γενικά ότι θα έχουμε τα πάντα ή τίποτα πρώτης Λισαβόνας μετά τη Λισαβόνας. Δούμε ε, ποιοι είναι οι φάκελοι όπου μπορούμε όντως να έχουμε ε, ένα αποτέλεσμα. Ωραία. Προτού δώσω το λόγο στον κύριο Διαζεμία θα ήθελα να πω για να αποφύγω παρανοήσεις ε, ότι όπως είπε η κυρία Φαγιόν ε, που ζήτησε μία ταχεία υιοθέτηση υπάρχουν τέσσερις διαδικασίες όπου είναι ακατανόητο γιατί θα πρέπει να υιοθετηθούν στο συμβουλιο πρώτης πρώτης 1ης δεκεμβριου Ζητώ λοιπόν το Συμβούλιο να μου εξηγήσει γιατί. Η κυρία δίας Ο κύριος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος αλλά σαφής. Τώρα σχετικά με τα τέσσερα αιτήματα της Europol, το Συμβούλιο της 26 Απριλίου, το οποίο ήμουν εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Σώμα, αποφασίστηκε σύμφωνα με την άποψη του Κοινοβουλίου και όχι με την συνδιαλλαγή, στην απόφαση. Ε, κατά άποψή λοιπόν το Συμβούλιο υιοθέτησε μόνο το 20% των ε, συστάσεών μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε τώρα σε ένα νομικό πλαίσιο εντελώς διαφορετικό. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα πλαίσιο που μας δεσμεύει, αρχή μας δεσμεύει η συναπόφαση με την ε, ε, από την έναρξη της ισχύου διαδικασία τη συνθήκη της Αγώνα από την 1η Δεκεμβρίου. Λοιπόν, έχουμε τώρα ένα ζήτημα που αφορά την ε, ρυθμίσει ανάπτυξη, ε, ρυθμίσει εμπιστευτικότητα και κανόνων που διέπουν τη σχέση της Europol με τους εταίρους της στο θέμα ανταλλαγής πληροφοριών και δι χαρακτηρισμένων στοιχείων. Κάτι το οποίο δεν είναι ίσονο σημασία. Κατά νέο μου λοιπόν είναι παράλογο ενώ πρόκειται να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αστυνομίας ε, υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο σε, με, που θα προβλέπεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό και με κοινοτικούς υπαλλήλους στελεχωμένοι εάν εδώ για 15 μέρες μας αφαρείται τη δυνατότητα να πούμε και να προωθήσουμε τα κοινοβουλευτικά και νομικά μας επιχειρήματα τώρα με τη θέση τη αγώνας. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφύγει τις ευθύνες του Σύμφωνα με τη λογική λοιπόν για το την υπηρεσία αυτή της Ευρωπαϊκής Αστυνομία, το Συμβούλιο πρέπει να συναφασίσει με το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν πρέπει μόνο να εκφράσει γνώμη, πρέπει να εισακουστεί. Εγώ πρόεδρε αναγγέλλω πως οι τέσσερις συγγυητές ε, επί των τεσσάρων εκθέσεων θα υποβάλουν μια τροπολογία για όλα αυτά και ζητώ από το Συμβούλιο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμά του προκειμένου να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να υλοποιήσουμε την, να πραγματοποιήσουμε όλη αυτή την έκθεση σίγουρα με τη Σύγκλη Λισαβόνας. Πρέπει να δώσω το λόγο τον κύριο Κύρκοπ, ο κύριο Γκούτ, διευθυντής του γραφείου παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας αλλά το λόγο ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει δεν είναι ζήτημα γένειας απέναντι στο πρόσωπό του ο κύριος Κύρκοπ θα είναι ο τελευταίος ομιλητής και αν κάποιος άλλος έχει κάνει αυτό ζήτημα να δείξει θα ολοκληρώνουμε τον κατάλογο και θα δώσουμε το λόγο στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ακούσαμε τους νομικούς. Μα ανησυχεί το γεγονός, με ανησυχούσε το γεγονό ότι διάφορα σημαντικά πράγματα έτσι τα πιέζουμε, περνάνε έτσι πολύ ταχαίω από την Επιτροπή μα, ακόμα και το δικό μου θέμα ε, που αφορά τα εγκληματολογικά εργαστήρια που θα έπρεπε να συζητηθεί σήμερα. Ε, έγραψα στην νομική υπηρεσία ε, για το θέμα τη νομική βάση που πρόκειται να αλλάξει το Συμβούλιο. Και έγραψα και στο Συμβούλιο και ζήτησα να μου απαντήσει για το θέμα τη νομική βάση, που είναι πολύ σημαντικό στατικό αν θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θέλω μια απάντηση σήμερα. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι προφανώς είναι σημαντικό θέμα, θα πρέπει να καθορίσουμε τη συνολική βάση με τη Λισαβόνα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει χρονική πίεση κτλ. Και, και εγώ δεν θα είμαι σε θέση να συνεχίζω, γιατί δεν έχω καθόλου απαντήσεις από τους νομικούς για το θέμα που με απασχολεί η νομική βάση δηλαδή. Νομίζω ότι θα αντιμετώπισα μεγάλη πίεση. Υπάρχουν διάφορε εκθέσει, όπω και η δική μου, ε, που δεν θα διεκπαιρεωθούν. Και τα θέματα που θέτουμε με αυτέ τι εκθέσει είναι πάρα πολύ ζωτική σημασία. Όλα ε, οφείλονται στην πίεση στην οποία υποβαλλόμαστε. Ε, και μα πιέζουν να ε, τσεκάρουμε όσο δυνατόν περισσότερα κουτιά, α πούμε, κουτάκια πριν περάσουμε στη Λισαβόνα. Δεν μου αρέσει αυτή η πίεση. Δεν έχω καμία απάντηση από την νομική υπηρεσία ή από την νομική κοινότητα προ την οποία απευθύνθηκα. Και αν και εφόσον δεν έχω, είμαι πραγματικά σε δύσκολη θέση. Τι να κάνω. Ε, θέσατε ένα θέμα λοιπόν σαφώ προ την νομική υπηρεσία η οποία εξακολουθεί να εκπροσωπείται. Ο κύριο Γκάτ νομίζω θα μα βοηθήσει για να το κλείσουμε αυτό το θέμα σε λίγα λεπτά. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν η νομική υπηρεσία να απαντήσει στο τελευταίο θέμα και συνεχεία Στρέφουμε προς τη γραμματεία και θέλω να πω ότι αύριο, πριν τη συνεδρίαση των συντονιστών, θα πρέπει να υπάρχει ένα λεπτομερή κατάλογο, όπω προτείνει και ο κ. Μπουσουτήλ, με όλε τι εκκρεμεί διαδικασίε και την νομικό, νομική κατάσταση της επιπτώσης στο βαθμό του επίγοντα χαρακτήρα. Και θα ήθελα μετά την συνεδρία των συντονιστών να πούμε ποια είναι η θέση μας για κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες και να ζητήσουμε μία απάντηση, κατά προτίμηση γραπτή, από το Συμβούλιο, καθώς και μια εξήγηση γιατί κάποιες ε, διαδικασίες είναι τόσο πια επίγουσες που θα πρέπει ντε και καλά να υιοθετηθούν πριν τη θέση σε ισχύ της Λισαβόνας. Γιατί νομίζω ότι μας το οφείλει το Κοινοβούλιο, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά το οφείλει και στους Ευρωπαίους πολίτες. Το ΛΙΚ το ξαναλέω αυτό. Ε, κλείνω λοιπόν. Θα κλείσουμε τώρα με την ε, απάντηση της νομικής υπηρεσίας και με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά από από αυτό που με επικραμματεί, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε στις 4.30. Αλλά θα μπορούσα να σα παρουσιάσω και τώρα τη γνωμοδότησή μου προφορικά, εάν το επιθυμεί η Επιτροπή. Κύριε Κέρκο, θέλετε μια απάντηση για το θέμα σα ή τη στιγμή που θα θέσουμε που θα τεθεί το δικό σας θέμα. Ε, δεν θέλω να κρατήσω εδώ τους δικηγόρους, γιατί ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θα ήθελα μια σύντομη απάντηση τώρα, θα με βοηθούσε πολύ. Πολύ ωραία. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να απαντήσετε σύντομα. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά όπως ξέρετε, εγώ διαθέτω το χρόνο μου δωρεάν για την Επιτροπή τη δική σας. Ε, ο κύριος Λόπες έθεσε δύο ερωτήματα για την νομική βάση της, πρότα... πρότασης πλαίσιο για την ε, πιστοποίηση των ε, εγκληματολογικών εργαστηρίων. Είναι σωστό να αναφέρουμε το άρθρο 31 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό, 31, αναφέρει ότι η Ένωση μπορεί να αναλάβει ε, κοινή δράση για την ε, δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα. Δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα, το τονίζω. Ε, η προτινόμενη απόφαση πλαίσιο, από ό,τι βλέπουμε, δεν καλύπτει την δικαστική συνεργασία, την αστυνομική συνεργασία. Και το άρθρο 5.2 της πρότασης ε, ρητά λέει ότι η απόφαση πλαίσιο δεν επηρεάζει τους εθνικούς κανόνες για την δικαστική αξιολόγηση. Επομένως, η διαγραφή του άρθρου 31 νομίζω ότι δικαιολογείται. Το δεύτερο ερώτημα είναι πιο δύσκολο να απαντηθεί. Και ο κύριος Λόπες ε, στο γράμμα του λέει ότι η απόφαση πλαίσιο επίσης αριθμίσει και τις δραστηριότητε και των δημόσιων αρχών και των εταιριών ε, ιδιωτικού χαρακτήρα που ε, ασχολούνται με εγκληματολογικές υποθέσεις. Μιλάμε για υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 51, 50 συγγνώμη, της συνθήκης ΕΚΑ. Και αν ναι, τότε εντάσσονται στην αρχή και στο πεδίο της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρώτου πυλώνα και επομένως ε, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα υπό τον τρίτο πυλώνα. Άρθρο 47 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ε, είπε το... Ερμήνευσε και το δικαστήριο με βάση την ε, πράξη για τα μικρά όπλα. Λοιπόν, ο ε, ορισμό του άρθρου 50 είναι πολύ ευρύ και περιλαμβάνει όλε τι υπηρεσίε που κανονικά παρέχονται επαμοιβή. Επομένω, αν η ιδιωτική εταιρεία κάνει ε, εργαστηριακέ δραστηριότητε για την αστυνομία, προφανώ τι κάνει επαμοιβή. Δίνει δηλαδή μια υπηρεσία. Τώρα, το Συμβούλιο θα πρέπει να δείξει ή δεν υπάρχουν ιδιωτικέ εταιρείε που δίνουν υπηρεσία ή αν την τη δίνουν αυτή την υπηρεσία, τότε ε, δεν την κάνουν επανειδή. Και δεν είναι απλό αυτό. Εάν οι εργαστηριακές υπηρεσίες θεωρούνται ε, υπηρεσία, τότε μπορεί να εντάσσονται στα πλαίσια μιας παρέκκλησης που προβλέπει το άρθρο 45 και 55 της συνθήκης ΕΚΑ. Αυτή η παρέκκληση λέει ότι οι δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται ακόμα και περιστασιακά με την ε, με τις δραστηριότητες των δημοσίων αρχών αποκλείονται. Και η νομολογία του δικαστηρίου ερμηνεύει αυτόν τον αποκλεισμό πολύ ε, περιοριστικά. Ε, το δικαστήριο λέει ότι αυτές οι δραστηριότητες των εργαστηρίων δεν εντάσσονται στην ε, παρέκκληση για τις επίσημες δραστηριότητες. Ε, τώρα, αυτές οι δραστηριότητες που λέει η απόφαση πλαίσιο είναι ίσως δευτερεύουσες για, την, για τις διοκτικές αρχές. Καταληκτικά λοιπόν. Εάν ε, το Συμβούλιο δεν μας δείξει ότι οι υπηρεσίες αυτών των εργαστηρίων, όπως ε, προβλέπονται από την απόφαση πλαίσιο, δεν εντάσσονται στο άρθρο 50, τότε θεωρούμε ότι δεν μπορούν να ρυθμιστούν με βάση τα μέτρα του τρίτου πυλώνα. Αυτό τι σημαίνει. Ε, ότι το θέμα βγαίνει από την μέση διάταξη. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς οι μη ειδικοί. Μάλιστα. Ε, θα, ήθελα, ε, θα ήθελα να με χρεώσετε τότε ε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο που το ΦΠΑ μας θα είναι 15%. Ευχαριστώ την νομική υπηρεσία, τη Σουηδική Προεδρία. Ο κύριος Γκουτς, πού είναι? Συγγνώμη, μπορείτε να αποχωρήσετε ησύχω τη αιθούση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την συνεδρίασή μα. Κυρία Αλφάνο, έχετε ένα, ένα διαδικαστικό. Ναι, Πρόεδρε. Αφορά στις διαδικασίες που θα συναντήσουμε μπροστά μας. Το θέμα του δικτύου για την πρόληψη του εγκλήματος διακόπτη προς... Ε, θα σας διακόψω διότι τη συζήτηση την κάναμε σχετικά με τις εκκρεμούσες διαδικασίες. Θέλετε να το συζητήσουμε τώρα το θέμα ή μπορούμε να το συζητήσουμε στο πλαίσιο των συντονιστών. Ναι, μπορούμε να το εξετάσουμε αύριο το πρωί, παρατηρή κυρία Αλφάνο. Κύριε Γκούρτσου, ευχαριστώ για την επικία σας και την υπομονή σας. Θα θέλαμε να ακούσουμε την παρουσίαση της σας εκθέσεως. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο σας δίνω μία νέα έκθεση αλλά όχι μία νέα συνθήκη τη Λισαβόνα, γι' αυτό και κατανοώ τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερος Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι διότι σήμερα ε, ουσιαστικά μπορώ να σας παρουσιάσω την επίλυση πολλών προβλημάτων μας ε, για την παρακολούθηση ναρκωτικών στην Ευρώπη για την κατάσταση εις ε, τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ε, Κροατία, την Τουρκία και άλλες γειτονικές χώρες. Κατά αυτόν τον τρόπο ε, θα δείτε στο διαδίκτυο ότι υπάρχουν τα στοιχεία μας διότι δημοσιεύουμε διάφορα θέματα ενδιαφέροντος και μία ανάλυση της πρακτικής για μαζικά εγκλήματα τοξικομανών, ε, μία έκθεση για τα διάφορα ναρκωτικά και για μία έκθεση για τα συνθήματα συνθετικά παράγωγα κάναβης. Μπορώ να σας αναφέρω μόνο τα τηλεγραφικά ορισμένα θέματα, αλλά αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που θα θίξω και θα δείτε ότι η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Προτού τώρα προχωρήσω στο περιεχόμενο της εκθέσεως θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεσή μας βασίζεται σε ανταλλαγές με όλους τους εμπειρογνώμονες της Ευρώπης. Και γι' αυτό όπως και κάθε χρόνο κάνουμε μία επισκόπηση της κατάστασης σε όλες τις χώρες και αξιολογούμε και την εθνική ε, εικόνα του προβλήματος για κάθε χώρα. Ε, εδώ θα ήθελα εδώ να αναφέρω την ε, εργασία του δικτύου για τα σημεία επαφής. Ξέρω ότι υπάρχουν θέματα ε, τα οποία μας ενδιαφέρουν πολύ και από αυτά που σας είπα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ορισμένα θέματα επιβεβαιώνουν τώρα και μπορούμε συνολικά να πούμε ότι η κατανάλωση των ναρκωτικών στην Ευρώπη είναι σε υψηλό επίπεδο αλλά αρκετά σταθερή. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε για μια βελτίωση της κατανάλωσης ηρωίνης και κοκαίνης που μας απασχολούν ιδιαιτέρως γιατί ε, έχουν μεγάλες δυνατότητες να επηρεάσουν αρνητικά την εθνική ασφάλεια και ε, την ε, τις ελευθερίες. Θα ήθελα να αναφερθώ στην κοκαίνη. Τέσσερα εκατομμύρια ενήλικες έχουν καταναλώσει αυτό το ναρκωτικό πέρυσι στην Ευρώπη ε, και ε, προσπαθούμε ε, να εξετάσουμε ε, το, τις δυνατότητες της κοκαίνης που επεκτείνονται σε όλες τις Ευρώπης και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει παραγωγή κοκαίνης σε χώρες Ανατολικής Ευρώπης και ότι διακινούνται όλο και περισσότερο στα νυχτερινά κέντρα της περιοχής αυτής. Μαζί με την Ευρωπόλη, λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε μία κοινή αξιολόγηση της αγοράς της κοκαίνης στις διάφορες πτυχές της. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, Νορβηγία υπάρχουν 1,5 ε, εκατομμύριο προβληματικοί καταναλωτές εκ των οποίων οι περισσότεροι καταναλώνουν ηρωίνη. Δεν μιλάμε για επιδημία αλλά υπάρχει αύξηση κατανάλωσης της ηρωίνης άρα το πρόβλημα οξύνεται και δεν μειώνεται. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει και αύξηση αιτήσεων θεραπείας αλλά και θανάτων από τα ναρκωτικά αυτά ο αριθμός της διαθέσεως η ηρωίνη στην Ευρώπη έχει αυξηθεί και η διακίνηση ε, ε, ε, στην Τουρκία από 2,7 εκατομμύρια έφτασε στο 5 στα 13 εκατομμύρια. Αν λοιπόν αξιολογήσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες πρέπει να πούμε ότι η ηρωίνη δεν αποτελεί πρόβλημα του παρελθόντος και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις βλάβες και ε, να αναγνωρίζουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όταν υπάρχει κατανάλωση ηρωίνης στους νέους ή σε ε, ε, επισφαλείς ομάδες. Υπάρχει επίσης μεγάλη ζήτηση για κάναβη. Ε, διότι πολλά εκατομμύρια ε, των συνανθρώπων μας έχουν ε, χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους κάναβη, δηλαδή το 1 τέταρτο του ενήλικα πληθυσμού. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι οι νέες τάσεις μας οδηγούν σε κάποια αισιοδοξία διότι ενώ στη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 είχαμε μία αύξηση ε, της ε, ε, της καταναλώσεως βλέπουμε ότι τώρα μειώνεται η προσέλκυση ιδίως των νέων και ε, εξετάσαμε ιδιαίτερα την κατανάλωση από παιδιά σε σχολική ηλικία στην Ευρώπη ε, και παρόλο που βλέπουμε μία σχετική αύξηση υπάρχει μία σταθερή εξέλιξη και μείωση σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη. Την ίδια μείωση βλέπουμε και στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Αυστραλία. Όταν μιλούμε λοιπόν για κατανάλωση της κάναβης πρέπει ε, να εξετάσουμε ε, τις τάσεις και οι τάσεις αυτές ε, δεν συνάδουν με την ε, εικόνα που περιέγραψα διότι 2,5% των Ευρωπαίων περίπου 3 εκατομμύρια νέων καταναλώνουν καθημερινά κάναβη και αποτελούν μια επικίνδυνη ομάδα όσον αφορά δε την ζήτηση η οποία έχει σταθεροποιηθεί δεν ξέρουμε αν έχει σταθεροποιηθεί σταθεροποιηθεί λόγω έλλειψης προσφοράς ή σταθεροποίηση της ζήτησης θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν προληπτικά μέτρα πολύ πιο σημαντικά και καινοτόμες διαδικασίες διότι στους νέους παραδείγματος χάρη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επεμβούμε διότι οι νέοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πληροφόρηση και για ανταλλαγή μηνυμάτων και εδώ έχω αναφέρει μόνο τα παραδείγματα παραδοσιακά προβλήματα της Ευρώπης αλλά τώρα θέλω να στραφώ προς το ερώτημα των επιπτώσεων για την πολιτική διότι συνήθως μιλώ με τους ειδικού για τη θεραπεία και εκεί λέγω ότι τα άτομα τα οποία καταναλώνουν μόνο μία ουσία αποτελούν μειοψηφία πλέον. Δηλαδή υπάρχουν ένα σωρό ψυχοφάρμακα τα οποία καταναλώνουν συνδυασμένα πολλοί από αυτούς τους νέους και αυτό αποτελεί μία νέα πρόκληση την οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Όσον αφορά την πολιτική μας προοπτική διαπιστώνουμε ότι ο συνδυασμός ο ινοπνεύματος και των ναρκωτικών αποτελεί μια νέα κατάσταση την οποία πρέπει να σπάσουμε. Ε, και βλέπουμε ε, ότι ε, συγχρόνως υπάρχει κατάχρηση νοπνεύματος και συνδυασμός με, με κατανάλωση ναρκωτικών και γι' αυτό θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε και πάλι την απομάκρυνση από κατανάλωση μία μόνο και κλίση προς συνδυασμό πολλών ουσιών και ούτως ή άλλως τα ναρκωτικά είναι εμπορεύματα τα οποία ανταγωνίζονται και ατυχώς είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να επιλύσουμε εμείς. Θα ήθελα όμως να σας πω ποια είναι τα νέα συνθετικά ναρκωτικά που διαπιστώσαμε στην αγορά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες χημικές ουσίες και προσπάθειες οι οποίες προσπαθούν να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ελέγχου. ή μεταφεταμίνες παραδείγματος χάρη οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη και υπάρχει και μια ανησυχητική εξέλιξη διότι οι μεταφεταμίνες προσφέρουν όλο και περισσότερο στη Βόρειο Ευρώπη Ευρώπη όπου μέχρι στιγμής υπήρχαν μόνο αμφεταμίνες στην Σλοβακία και σε γειτονικέ χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατανάλωση της μεταμφεταμίνης έχει αυξηθεί καθώς και τα συμπαρατούμενα προβλήματα και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει εδώ μία, ένα ναρκωτικό το οποίο εύκολα παράγεται σε ένα γκαράζ και ε, μπορεί να διατεθεί ε, όλο και περισσότερο οπότε πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη. Η αλλαγή των ε, συνθήκων διαθέσεως ισχύει και για τις, ε, τα νέα δισκία ε, έκσταση διότι η MTA που ήταν η ουσία του έκσταση έχει αντικατασταθεί με το MCPP η οποία δεν υπόκειται σε κανένα έλεγχο στην Ευρώπη. Τώρα το εάν πρόκειται για μία προσωρινή αλλαγή ή για μία μόνιμη αλλαγή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τώρα και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε. Από πλευράς παρακολουθήσεως των ναρκωτικών επίσης να τονίσουμε Ευχαριστούμε ε, την, την ύπαρξη μίας αγοράς όπου δεν προσφέρονται ε, ουσίες ελέγχου. Αυτό δεν είναι νέο, αλλά το νέο είναι ότι παρισφρεί όλο και περισσότερο χρήση του διαδικτύου για την διάθεση προϊόντων με ψεύτικες ετικέτες και ε, μεγάλη ταχύτητα με την οποία η αγορά αυτά, αυτή αντιδρά εφόσον ληφθούν μέτρα ελέγχου. Το Spice π.χ. Ένα προϊόν το οποίο περιέχει συνθετική κάναβη ε, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, ε, μάλλον διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε συνεργασία με την Europol και εδώ πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο διατίθεται στην Ευρώπη αλλά κατασκευάζεται στην εργασία γιατί είναι πιο φτηνό και ε, αποβλέπει σε μεγάλες ε, τάξεις καταναλωτών οι οποίοι ενδιαφερόντουσαν για την κάναβη και προσφέρεται σε πολύ ενδιαφέρουσες συσκευασίες μας δίνει μία πρόγευση του τι μας περιμένει στο μέλλον σχετικά με τους ε, μηχανισμούς ελέγχου των ναρκωτικών και γι' αυτό ε, θα πρέπει να παρακολουθούμε τις ε, νέες εξελίξεις της αγοράς. Πρέπει να σας πω ότι με την έκθεση αυτή προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε μία επισκόπηση των προβλημάτων των ναρκωτικών στην Ευρώπη και των μέτρων τα οποία σκοπεύουμε να, λάβει, ε, να λάβουμε και ε, θεωρούμε ότι πρέπει να προέχει η ε, επιστημονική αντιμετώπιση και όχι η κομματική ή συγκινησιακή ε, αντιμετώπιση. Πιστεύω λοιπόν ότι με την εργασία μας αυτή θα μπορέσουμε ε, να ε, προκαλέσουμε μία πολιτική συζήτηση κατά τρόπον ώστε να σας δώσουμε σε εσά που παίρνετε τις πολιτικές αποφάσεις τη δυνατότητα να λάβετε τα δέοντα μέτρα. Η έκθεση την οποία βρήκατε σήμερα είτε ε, χθε δεν θα πρέπει να κοινοποιηθεί μέχρι αύριο το πρωί στις 10 που θα διατεθεί στον τύπο. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ε, ότι κατάλαβα όλα τα μέλη έχουν λάβει ένα αντίγραφο, εγώ λαμβάνω τώρα. Φυσικά είναι μια συζήτηση η οποία προκαλεί πολλές αντιδράσεις, ε, γι' αυτό όμως είμαστε εδώ οι πολιτικοί. Λοιπόν, αν ε, όποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Κύριε Γιακουλίνο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κότσο για την ε, αναλυτική και σαφή παρουσίαση των δραστηριοτήτων ε, του τρέχοντος έτους. Έχω να κάνω κάποια σχόλια και κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Γκότς αναφέρθηκε στην εξέλιξη της κατανάλωσης ναρκωτικών που είναι ιδιαίτερα υψηλό αλλά και φύστερη διακυμάνση συνδέεται με μια αναπτυσσόμενη αγορά μας ανεφέρει για νέα ε, ναρκωτικά τα οποία χρησιμοποιούν για την ε, πώληση και την προφορική και αναφέρθηκε επίσης ε, σε δύο ζητήματα σημαντικά, την πρόληψη και την κουλτούρα της πρόληψης που θα πρέπει να συνδυαστεί κατά όψή μου με μια ε, συμμετοχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και μας είπε και κάτι άλλο το εξίσου σημαντικό που συνδέεται με τις εξελίξεις αυτής ε, της ε, αυξανόμενης διάδοσης και κατανάλωση ναρκωτικών που συνδέεται και με, τα, με το κατανάλωση αλκοόλ. Η πρόσβαση στα ελαφρά ναρκωτικά και στο αλκοόλ οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή την ε, εγκληματικότητα πρέπει να το αντιμετωπίσει το θέμα, πολλές πολλά σοφρονιστικά ιδρύματα στην Ευρώπη έχουν ε, ένα 5% του πληθυσμού τους που, ατόμων που κρατούνται για λόγους ναρκωτικών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν προληπτικά μέτρα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, σχέδια τα οποία έχουν προωθηθεί μέσω των επιχειρησιακών ομάδων και δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επεξεργάζονται τις πληροφορίες που μας προσφέρει το παρατηρητήριο. Δύο ερωτήσεις τις ε, προσεχείς μέρες. Πρόκειται να εγκριθούν ε, κάποιες ε, αποφάσεις, ε, κατευθύνσεις κλπ. Θα αναγνωρίζω αν αυτές οι κατευθύνσεις θα βασιστούν στα όσα μας είπατε, αν τα προγράμματα αυτά είναι σύμφωνα με τις προσπάθειες ε, ανάκτησης ε, των ε, ναρκωμανών, των τοξικομανών και αν υπάρχει μια πραγματική συνεργασία, όπως και θα ήταν χρήσιμο, κάτι τέτοιο, με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Υπουργεία Υγείας, διότι <coughs> υπάρχουν κάποιες σημαντικές εμπειρίες οι οποίες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να δείξουμε λοιπόν να πρέπει την αμοιβαιότητα για να προχωρήσουμε σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Σούγκο. Ευχαριστώ. Θα... Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας θέσω διάφορα ερωτήματα. Καταρχάς, ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Υπάρχει ισότητα ευκαιριών πραγματικά σε ό,τι αφορά την τοξικομανία ε, στις φυλακές. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την κατάσταση στη Ρουμανία. Η Ρουμανία δεν είναι μόνο χώρα διαμετακόμισης των ναρκωτικών, αλλά και χώρα κατανάλωσης, ιδίως κοκαίνης. Και έχω και ένα τρίτο ερώτημα. Δεν έχετε μετάφραση? Υπάρχει πρόβλημα με τη μετάφραση? από κάποια γλώσσα. Εγώ άκουγα τα αγγλικά, αλλά τα γερμανικά είχαν πρόβλημα. Γερμανική καμπίνα. Ε, τι κάνει η γερμανική καμπίνα. It's okay now. Εντάξει, ακούγεται τώρα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Ζητώ συγγνώμη. Μπορώ να το πω και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και στα γερμανικά αλλά και μια και η ουγγρική γλώσσα είναι απαγορευμένη σε ορισμένε χώρε, θα ήθελα να τη χρησιμοποιήσω. Όχι, και εμεί θέλουμε να την ακούσουμε, λέει η Πρόεδρο αυτή τη γλώσσα. Να επαναλάβω λοιπόν. Πολύ ωραία. Το πρώτο ερώτημα ήταν το εξή. Υπάρχει ισότητα ευκαιριών στις φυλακέ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ήδη, ε, ιδίως και έπειτα, Ποιε είναι ποιες είναι οι πιο προκλήσει τη της τη Ανατολική Ευρώπη, Η Ρουμανία, α πούμε, δεν είναι μόνο χώρα διαμετακόμιση των ναρκωτικών, ε, αλλά και κατανάλωση, ιδίω ε, κοκαίνης. Τρίτο ερώτημα. Τρίτο ερώτημα αφορά ένα πολύ σημαντικό εστιακό σημείο. Τα εστιακά σημεία, μάλλον. Τα εστιακά σημεία είναι τα ίδια ε, στη Ρουμανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ. Ρενάτα Βέμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ, κύριε Γκότς, για την ε, παρουσίασή σας και για τη δουλειά που κάνατε. Ομολογώ ότι δεν είχα το χρόνο να εξετάσω την έκθεσή σας, γιατί μόλις την έλαβα. Έχω τρεις ερωτήσεις, σύντομες. Μπορεί να απαντώνται, να δίνονται οι απαντήσεις στην έκθεση, αλλά θέλω να τις θέσω παρόλα αυτά προφορικά. Αναφέρατε ότι η κάναβης ε, είναι λιγότερο δημοφιλής ε, τώρα. Ε, η ερώτησή μου είναι, αντικαταστάθηκε με κάτι άλλο, μια άλλη ναρκωτική ουσία πιο δυνατή ίσως. Δεύτερη ερώτηση. η οδός της κοκαίνης. Είναι αλήθεια ότι ξεκινάει από Λατινική Αμερική, Δυτική Αφρική και εν συνεχεία Ευρώπη. Αυτή είναι, αυτός είναι ο δρόμος, αυτός είναι ο κύκλος. Και τρίτο ερώτημα. Το κέντρο σας έκανε ή θα κάνει μία ανάλυση της κατάστασης σε χώρες όπου η κατανάλωση ε, λαφρών ναρκωτικών έχει αποποινικοποιηθεί. Μιλάω βοήθεια προς τους χρήστες, ε, θεραπείες που υπάρχουν στη διάθεσή τους κτλ. Πριν δώσω το λόγο στον Νίκ, έχω και άλλους τρεις ομιλητές στον κατάλογό μου. Κύριε Γκουτς, θέλετε να απαντήσετε, να ακούσουμε πρώτα όλες τις ερωτήσεις και μετά απαντάτε. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διασταυρούμενη, η πολλαπλή χρήση ναρκωτικών είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί, είπατε. Είπατε ότι η νοποσία μαζί με τη χρήση ναρκωτικών είναι κάτω συνήθες θα ήθελα να σας ζητήσω ε, ποιες είναι οι πολιτικές ελέγχου. Αυτά τα φαινόμενα χρειάζεται μια νέα προσέγγιση ε, ως προς τον έλεγχο, δηλαδή κάποιες πολιτικές ελέγχου και κάτι που συνδέεται με αυτό. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να προωθήσουμε, κάποιες πολιτικές ας πούμε, που να βασίζονται σε κάποιες αποδείξεις, σε κάποιες ενδείξεις ας πούμε, που έχουμε. Παραδείγματο χάρη, ο βασικός σύμβουλος ε, του κύριου ε, συμβουλευτικού φορέα για τα ναρκωτικά μόλις απολύθηκε από τον Υπουργό στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ίσως υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην προσέγγιση αυτών που θέλουν να προωθήσουν την ποινικοποίηση, ε, τη δίωξη, εν και αυτούς που έχουν άλλη προσέγγιση Ευχαριστώ. Όλοι είσαστε πολύ λακωνικοί σήμερα. Πολύ καλό είναι αυτό. Κύριε Μπρόγκς, ο κύριος Μπρόνξ. Οι δραστηριότητε τη αστυνομία στο Ηνωμένο ε, Βασίλειο αντίον των Λαθρεμπόρων ναρκωτικών επικεντρώνονται σε εκείνου του λαθρέμπορου που είναι και χρήστε. Δηλαδή ε, στου μικρού, α πούμε, ε, της αλυσίδας. Και είναι απρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε του λαθρεμπόρου που δεν είναι χρήστε. Γιατί αυτοί, ε, ξέρετε ότι οι αστυνομικοί ζουν σε επικίνδυνες ε, περιοχές. Ε, γράφονται πηχιαίοι τίτλοι βέβαια όταν ε, πιάνουμε τέτοιους ε, χρήστες που βρίσκονται κάτω-κάτω στην αλυσίδα, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι τιμές και δεν μειώνεται η χρήση ναρκωτικών. Απλώς αυξάνονται οι τιμές, επομένως ε, γίνονται περισσότερες ληστείες, ε, πάμε περισσότερα αυτοκίνητα κτλ. Με αυτή την κατάσταση. Τώρα από τη ζήτηση εκεί δεν εστιάζουμε, δεν υπάρχει προσοχή. Οι dealer ε, που είναι και χρήστες μπαίνουν φυλακή για σύντομο χρονικό διάστημα όταν απελευθερώνονται, δεν έχουν υποστήριξη. Ακόμα και αν φύγουν από εκεί, από το κύκλωμα ας πούμε, ξαναμπαίνουν στις φυλακές σε 24 ώρες και γενικά στο κύκλωμα. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε ε, ρεαλιστές. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε με τοπική επίθεση ε, και δεν έχει νόημα να απαντούμε έτσι, να αντιμετωπίζουμε το θέμα ε, με πολύ συνετά, έτσι, να, να γδέρνουμε ας πούμε τις άκρες του προβλήματος, αλλά να μην το αντιμετωπίζουμε στην ουσία. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, γιατί συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κύριος Βέμπερ. Υπάρχουν συγκριτικά εμπειρικά δεδομένα που μας επιτρέπουν να συγκρίνουμε τα διάφορα συστήματα ε, νομιμοποίησης, απελευθέρωσης ή ποινικοποίησης των ναρκωτικών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Τα κράτη-μέλη συχνά δεν θέλουν να συγκρίνουν τις εμπειρίες τους. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του παρατηρητηρίου είναι ότι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις των εμπειριών μας, να δούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Αν θυμάμαι καλά, ε, είχε γραφτεί μια πρόσφατη έκθεση από ένα Αμερικανικό Ινστιτούτο που έλεγε ποιες είναι οι εμπειρίες ε, από ποινικοποίηση των ναρκωτικών στην Πορτογαλία. Ε, οι επιπτώσεις ήταν πάρα πολύ θετικές για τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό καλό είναι να δούμε ποιες είναι οι διάφορες επιπτώσεις και ποια είναι τα διάφορα μοντέλα. Ποιε είναι οι διάφορε επιπτώσει λοιπόν των ε, συστημάτων ε, στη δημόσια υγεία. Τελευταίο ομιλητή είναι η κυρία Αλφάνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Γκότ ε, διότι η έκθεση που μας ε, διαβίβασε είναι πολύ αναλυτική, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά την περιγραφή της κατανάλωσης των ε, διαφόρων ουσιών και εγώ ασχολήθηκα ιδιαίτερα με αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Η ροήνη κοκαίνη δεν δείχνουν σημάδια μείωσης ε, στην κατανάλωση. Είδα επίσης ότι Αναφέρθηκε και το πρόγραμμα δράση ε, τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσεχή τριετία 2009-2012, ο ρόλο τη ε, κοινωνία των πολιτών και ήθελα να γνωρίζω Πώ ε, φαντάζεται το παρατηρητήριο τον ρόλο τη κοινωνία των πολιτών και την ευαισθητοποίηση στα σχολεία, δηλαδή μια διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων και των λιγότερων νέων. Τώρα, κάτι σε με αυτά που είπε η κυρία Βέμπερ, αυτό το εμπόριο των ναρκωτικών σε ε, μεγάλες δόσεις, ε, συναφερθήκατε σε κάποια εμπορία, έχουν ε, έχει εντοπιστεί ο ρόλος του οργανωμένου εγκλήματος στη διακίνηση αυτών των ε, ουσιών αλλά νομίζω ότι επειδή δεν είχα το χρόνο έτσι καλώς να το διαβάσω όλο το κείμενο, το διάτρεξα απλά, θα ήθελα να γνωρίζω τα ε, εγκλήματα τα οποία έχουν σχέση με την κατανάλωση ναρκωτικών και στην χώρα μου είχαμε τραγικά γεγονότα διότι υπήρξε πολύ ψηλό αριθμό εγκλημάτων και αξιόπινων πράξεων που συνδέθηκαν με την κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ. Ε, ποια θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή να είναι η απάντηση όχι μόνο σε ποινικό επίπεδο αλλά και σε θέμα ε, αστυνόμευσης ε, στη χώρα μου τα τελευταία χρόνια, ειδικά τον τελευταίο έτος, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε ποινικό επίπεδο, αλλά οι αστυνομικές δυνάμεις μπόρεσαν να δράσουν πιο, πιο προσεκτικά, πιο συγκεκριμένα αν θέλετε. Δηλαδή μπορούν ε, να αφαιρέσουν διπλώματα από οδηγού ή και σε σοβαρέ περιπτώσεις να κατασχέσουν και το αυτοκίνητο, το όχημα. Υπήρξαν, υπήρξε μια κατόμβη ατόμων που έχασαν τη ζωή τους ε, και αυτό οφείλεται στην ε, οδήγηση ατόμων που βρίσκονταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν εάν αυτό το θέμα εξετάστηκε και πω το παρατηρητήριο θα μπορούσε να λειτουργήσει και να μελετήσει καλύτερα αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις. Όχι. Και να θέσω εγώ την ερώτησή μου και να ζητήσω από τον κύριο Γκότς να απαντήσει. Αυτό ετέθηκε προηγούμενα σε άλλες χρονιές. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται δηλαδή ο ε, συσχετισμός ε, εθνικών στοιχείων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, κατασταλτικών πολιτικών, οι πολιτικές οι οποίες στοχεύουν στη μείωση, του, μείωση της ζημιάς, της βλάβης. Θεωρείται λοιπόν ότι και αναφέρομαι τώρα στην ε, παρτίση της κυρίας τι στοιχεία έχουμε, στις σχέσεις χάπτολα, τι στοιχεία έχουμε τώρα στην διάθεσή μας, διότι έχει ζητηθεί να υποληθεί έκθεση εμπειρογνωμόνων και υπήρχε μια περίπτωση όπου όταν υπέβαλαν τα πορίσματά τους αυτή η Επιτροπή διαλύθηκε και τα άτομα απολύθηκαν. θα ήταν νομίζω ιδιαίτερα χρήσιμο να ε, υπάρχει δυνατότητα σε βάθος λέει απόψεων μαζί σας όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη του εγγράφου και μια που απουσιάζει ο κ. Λόπεζ, ο, ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, να, να σας ρωτήσω αν είστε διατεθειμένος να έρθετε ε, σε μια ύστερη χρονική στιγμή για να σας θέσουμε ερωτήσεις, αφού φυσικά θα έχουμε μελετήσει σε βάθος την έκθεση σας. Έχετε λόγο. Ευχαριστώ. Αν θέλετε θα ξεκινήσω από το τέλος και θα προχωρήσω προς την αρχή. Θα συνεχίσω προς το παρόν αγγλικά. αν μου το ζητήσει η Επιτροπή μαζί με τους συναδέλφους μας να επανέλθουμε, ευχαριστώ, θα επανέλθουμε. Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με ε, τις ε, καταστατικές μεθόδους ε, και πρόληψη ε, βλάβης. Νομίζω το σύστημα έχει εξελιχθεί τους τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να σας πω ότι αυτό το μέτρο μειώνει την, τις βλάβες ή έχουμε καταστολή. Υπάρχει και καταστολή και πρόληψη της βλάβης σε όλες τις χώρες και το θέμα είναι τι συμπεριλαμβάνεται στις πολιτικές απαντήσεις, αποφάσεις. Ουσιαστικά εμείς προσφέρουμε τους αριθμούς και από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα ιδεολογικά και άλλα. Όλα αυτά λοιπόν συνυπολογίζονται και γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε εδώ σαν γραφείο με τα κράτη-μέλη και αυτό είναι το βασικό θέμα έχουμε 20, 25, 25 ε, συνεδριάσεις τεχνικές αναέτος όπου συμφωνούμε με τα κράτη-μέλη για τους τρόπους συλλογής των στοιχείων, μεθοδολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα κράτη-μέλη, δηλαδή ε, έχουμε, συγκεντρώνουμε ό,τι ζητούμε και στη σωστή μορφή, αλλά πέραν αυτού είναι προφανώς ότι οι πέντε επιδημιολογικοί μας δείκτες οι οποίοι είχαν υποβληθεί στους αρχηγούς κρατών και αναφέρονται σε απόφαση που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο δεν έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει όμως και μία δυσκολία όταν μιλάτε για εξέταση ε, στοιχείων του πληθυσμού δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται τακτικά σε όλες τις χώρες. Οπότε ε, όσον αφορά το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι προφανές ότι το έγκλημα αυτό είναι συνδυασμένο με την διακίνηση ναρκωτικών και αυτό αναφέρεται και στην διακίνηση ηρωίνης από το Αφγανιστάν και κοκαίνης από την Κολομβία αλλά και παραγωγή κάναβης στην Ευρώπη ή αλλού. Ε, είναι πιο περίπλοκο το θέμα. Ε, θα μπορούσατε να μην είχατε ρωτήσει και για την τρομοκρατία. Ευτυχώς δεν μου κάνετε τέτοιο ερώτημα. Ξέρουμε ότι πολλές από τις υπηρεσίες ε, θεραπείας προλήψεως ε, των βλαβών ανατίθενται σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και εκεί η κοινωνία των πολιτών έχει ένα ενεργό ρόλο Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ε, οι οποίες ε, υπησέρχονται αλλά ουσιαστικά το σκέλος αυτό αναλαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η οποία οργανώνει συνεδριάσεις μία-δύο φορές το χρόνο όπου συζητάνε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την κοινωνία των πολιτών. Όσον αφορά την αποποινικοποίηση, όπως ξέρετε ε, υπάρχουν σε όλες τις χώρες ε, τάσεις για αποποινικοποίηση και ε, ουσιαστικά είναι η φυσιολογική φυσιολογική αντίδραση από το κράτος. Ε, ένας ε, ε, δράστης στην πρώτη, ο ένας χρήστης την πρώτη φορά θα λάβει μία προειδοποίηση και μετά θα ακολουθήσουν τα άλλα μέτρα. Αλλά η κατάσταση είναι διαφορετική για την διακίνηση ναρκωτικών που στην Πορτογαλία ιδίως μία Αμερικάνικη εταιρεία λέγει ότι ε, στην Πορτογαλία ε, τα άτομα αυτά υποβάλλονται σε μία εξέταση από μία επιτροπή η οποία αποφασίζει εάν ε, τι θεραπεία θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται στην Πορτογαλία καμιά δεκαετία και έγιναν πολλά σχόλια ότι η Πορτογαλία θα γίνει το τοριστικός προορισμός για τους ναρκωμανούς αλλά αυτό βλέπουμε ότι δεν συνέβη αυτό μπορούμε να πούμε η κατάσταση στην Πορτογαλία δεν έχει ε, επιδεινωθεί δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και ε, <clears throat> δεν μπορούμε να σας δώσουμε άμεσες αποδείξεις και να σας πούμε ότι η πολιτική αυτή έχει αποδώσει αυτά τα αποτελέσματα απλώς θα μπορούμε να σας πούμε τι δεν έχει συμβεί. Μετά υπάρχει το, υπήρξε το ερώτημα ε, σχετικά με ε, ε, τα θέματα συνεργασίας με τις οργανώσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων όσον αφορά τις φυλακές γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία αποφυλακίζονται και δεν παρακολουθούνται. Είναι πολύ οξύ θέμα για τους χρήστες ηρωίνης διότι είναι ε, ακριβή η ε, προμήθεια ηρωίνης, ε, καταναλώνουν και μεγαλότερες... Ε, ποσότητες από ό,τι θα ήθελαν, έχουν δυνατότητα αν αποφυλακιστούν να ε, χρησιμοποιήσουν περις, μεγαλύτερες ποσότητες ηρωίνης και ε, έχουμε πολλές περιπτώσεις με υποτροπές αποφυλακιστέντων οι οποίοι είναι χρήστες ηρωίνης. Ε, ελέγχθησαν πολλά για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα σχολιάσω όμως γιατί κάθε κράτος έχει δικαίωμα να καταρτήσει τις επιτροπές του και δεν θα σχολιάσουμε εμείς στο σημείο αυτό. Όσο δεν αναφορά το θέμα ότι η δράση της αστυνομίας μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες περιοχές σε αύξηση της τιμής ισχύει σε τοπικό επίπεδο αλλά όχι αν μιλάτε για διεθνή διακίνηση όπου υπάρχουν υπάρχουν, ε, υπάρχουν κατασχέσεις ναρκωτικών που ήδη είχαν ε, προεξοφληθεί από τους διακινητές και ε, βλέπουμε ότι γενικά διεθνώς όλες οι παράνομες ουσίες έχουν μικρότερη κατανάλωση στην Ευρώπη, φθήνουσα κατανάλωση. Τώρα, Βεβαίως βασιζόμαστε σε αποδείξεις και προσπαθούμε να προσφέρουμε αποδείξεις για τη λήψη των αποφάσεών μας το ερώτημα του εάν υπάρχει ένταση ε, μεταξύ της κατασταλτικής διαδικασίας και της προλήψεως βλαβών όπως είπαμε με την βοήθεια των μεθόδων μπορέσαμε ε, να ε, αποσυμφορήσουμε το θέμα σημαντικά. Μία ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι εάν μειωθεί η χρήση κάναβης στους νέους αντικαθίσταται από κάτι άλλο δεν μπορώ να σας δώσω αριθμούς αλλά ενδεχομένως ε, μπορεί να ε, αντικατασταθεί ε, με κατάχρηση ινοπνεύματος και με άλλες ουσίες τις οποίες προανέφερα. Δηλαδή όλα αυτά τα νέα προϊόντα στην αγορά των συνθετικών ναρκωτικών που ε, διαφημίζουν ότι έχουν αποτέλεσμα σαν την κάναβη ε, και έχουμε δει ε, ότι ε, τα συνθετικά αυτά παράγωγα καναβής ε, ίσως έχουν εξεταστεί εργαστηριακά από τις φαρμακοβιομηχανίες αλλά ποτέ δεν έχουν παραχθεί βιομηχανικά. Η κάναβης ίσως δεν είναι πια τόσο δημοφιλή στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένε Πολιτείες και αλλού ίσως όπου δεν έχουμε προβεί σε μια ενδελεχή εξέταση και ενδεχομένως η πολιτική αυτή μπορεί να έχει ελαφρά επηρεάσει την κατάσταση αλλά ουσιαστικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με την καταπολέμηση του καπνίσματος διότι η κάναβης συνδυάζεται με το κάπνισμα και ξέρουμε ότι η πολιτική η καταπολέμηση του καπνίσματος είχε θετικό αποτέλεσμα και ορισμένα στοιχεία μας οδηγούν να πιστεύουμε ότι έτσι μειώνεται και η κατανάλωση κάναβης στους νέους. Όσον αφορά την κοκαίνη και τις ρίζες της, όντως η κοκαίνη ε, προέρχεται, ε, έρχεται στην Ευρώπη από διαφορετικές διαδρομές με κοντέινερ στην, ε, με εμπορευματοκιβώτια στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία ή αεροπορικά οι, μεγαλε, οι μεγάλες κατασχέσεις κοκαίνης στην Ευρώπη είναι ιδίως στην Ισπανία, στην Πορτογαλία λιγότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία. Περνά πολλές φορές από την ε, Δυτική Αφρική, δηλαδή είναι πάντοτε τα ίδια σημεία όπου υπάρχει ασταθής πολιτική κατάσταση που είναι πολύ πιο εύκολο να διέρθει κανείς από τις χώρες αυτές και ίσως ξέρετε ότι 7 κράτη-μέλη έχουν καταρτήσει μια ειδική οργάνωση για να καταπολεμήσουν την ε, ε, διακίνηση της κοκαΐνης ε, μέσω του Ατλαντικού με ανάλυση των θαλασσίων διαδρομών των ναρκωτικών και προσπαθούν να συνδυάσουν όλες τις πληροφορίες για να δουν ποιο πλοίο μπορεί να μεταφέρει κοκαίνη και άλλες ουσίες και οργανώνουν με το πολεμικό ναυτικό και την αστυνομία των, των πιο κοντινών χωρών τις κατασχέσεις και νομίζω ότι από αυτού έχει υπάρξει μεγάλη επιτυχία δεν θυμάμαι ακριβώς τους τους αριθμούς που επέτυχαν να κατασχέσουν τις ποσότητες δηλαδή πριν από 2-2,5 χρόνια αλλά ήταν σημαντικές. Όσον αφορά τις ανατολικές και δυτικές χώρες η κατάσταση είναι τέτοια ώστε στα νέα κράτη-μέλη στην κεντρική και Ανατολική Ευρώπη η κατανάλωση των παρανόμων ουσιών είναι συνήθως χαμηλή αλλά αυξάνεται τώρα και όντως όπως είπα και προηγουμένως έχουμε όλο και περισσότερες κατασχέσεις κοκαίνης στην, ε, σε ανατολικές χώρες οι οποίες δεν προορίζονται σε ανατολικές χώρες είναι απλούστατα μια διαφορετική μορφή διακίνησης δηλαδή μέσω Αφρικής ε, μέσω ε, άλλων χωρών και υπάρχουν δίκτυα τα οποία διέρχονται από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και άλλες παρεμφερείς χώρες. Υπάρχει μία αιστεία στην Ρουμανία η οποία ε, παρακολουθείται από την ε, ρωμανική... Ε, αστυνομία που παρακολουθεί τη διακίνηση ναρκωτικών ε, και ελπίζουμε ότι στη, η αιστεία ε, όπου ε, γίνεται αυτή η παρακολούθηση είναι στη Ρουμανία. Μιλήσαμε για ελαφρά φάρμακα, ελαφρά ναρκωτικά. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτών των όρων διότι είναι λιγότερο πρόβλημα κάποιος χρησιμοποιεί χρησιμοποιήσει κοκαίνη μια φορά στη ζωή του ή κάναβη κάθε μέρα. Οπότε ε, υπάρχουν διάφορες ε, μορφές ε, διάφορες μορφές κατανάλωσης και πρέπει να ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες μας διότι στην ιστοσελίδα μας έχουμε την πύλη των βελτίστων πρακτικών όπου μπορείτε να δείτε προγράμματα τα οποία έχουν επιτύχει σε ορισμένες χώρες και αξιολογούν διότι σε άλλες χώρες ίσως μπορεί να δώσουν την ευκαιρία να εφαρμοστούν παρεμφερία θέματα ε, με μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό η ιστοσελίδα αυτή ε, τη χάνει πάρα πολλών επισκέψεων ε, και αναφέρουμε και εκεί και μέτρα για κοινωνική ένταξη και πρότυπα για βέλτιστες πρακτικές. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Αν έχω παραλείψει καμία, παρακαλώ να μου το πείτε, αλλά και ευχαρίστω να επανέλθω στην Επιτροπή σας και να συζητήσουμε περαιτέρω το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε ως υπηρεσία διότι έχουμε δει ότι όλα αυτά τα χρόνια οι εκθέσεις σας είναι εξαιρετικής ποιότητας, μας παρέχεται σημαντική εμπειρογνωμοσύνη και οι συντονιστές της Επιτροπής μας θα εξετάσουν πιθανές ημερομηνίε για περαιτέρω συνάντηση για να συζητήσουμε εκτενέστερα την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιες ιδεολογικές διαφορές ε, σε αυτήν την Επιτροπή αναφορικά με τη χρήση των ναρκωτικών και ποιες οι πολιτικές θα ήταν πιο αποτελεσματικές, αλλά μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε επί ενός σημείου ότι είναι λυπηρό που ενώ ε, κερδίζονται πάρα πολλά χρήματα με τα ναρκωτικά θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία ξημών καλωσορίζει την εφαρμογή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Αυτή είναι μια κακή μέρα για τους ε, κακοποιούς εγκληματίες, διότι η Λισαβόνα μας επιτρέπει να ε, πλήξουμε και να καταπολεμήσουμε το έγκλημα πολύ πιο αποτελεσματικά. Μόλις συνειδητοποίησα ότι είμαστε απευθείας στο διαδίκτυο, εν Περνάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα προσφυλές ε, για την Επιτροπή μας. Ο εισηγητής είναι ο κύριος ε, Κάσουμαν. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα και σήμερα έχετε ενώπιόν σας ε, ε, ένα σχέδιο κοινοβουλευτικών ερωτήσεων ε, μετά από απαντήσεις που μας έδωσε η νομική υπηρεσία θα ήθελα να απευθύνω αυτές τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν και να ζητήσω από τον εισηγητή να εξηγήσει τις ερωτήσεις που πρόκειται να θέσουμε προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν αλλά αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι να εγκρίνουμε τις ερωτήσεις αυτές, να τις υιοθετήσουμε σήμερα στην Επιτροπή μας. Να υπενθυμίζω στα μέλη και θα ήθελα, θέλω να προδικάσω την παρουσίαση από τον κύριο Κάσμαν. Έχουμε εκφράσει ιδιαίτερα φιλόδοξες απόψεις. Και, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για φιλοδοξία όταν αναφερόμαστε στην διαφάνεια των εγγράφων κλπ. Τον Μάρτιο εγκρίναμε την θέση μας και ο Κάσουμερ θα μας ζητήσει σίγουρα να επιβεβαιώσουμε αυτήν την ε, άποψη. Παρακαλώ οι αποχωρούντες αιθούσει να αποχωρήσουν ησύχω. Είχαμε λοιπόν σε βάθος ζήτηση επί του θέματος στο σώμα μας, αλλά αυτό δεν έχει αντανακλαστεί από σοβαρές συζητήσει και σε βάθος στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Εν η νέα συνθήκη, την οποία συζητάγαμε προ λίγου, αλλά στο νομικό πλαίσιο εντό του οποίου δρούν τα θεσμικά όργανα και γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρξει μια σιγηρή πολιτική δέσμευση από πλευρά Κομισιών και Συμβουλίου να αναθεωρήσουν τους κανονισμούς τους, διότι αυτό δεν αφορά μόνο τι σχέσει μεταξύ των οργάνων, αλλά είναι αφορά τις σχέσεις που έχουμε εμείς ως θεσμικά όργανα με τους πολίτες μας και την διαφάνεια την οποία δικαιούνται να αποκτήσουν οι πολίτες μας. Να ζητήσω λοιπόν από τον Μάικλ Κάσμα να λάβει το λόγο και μετά το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα σχολιάσουν και θα ανοίξει η συζήτηση στην Επιτροπή. Μάικλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. με την έξοδο παρατήρησα ότι οι εξερχόμενοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα νομικά ζητήματα και για την πρόσβαση στα έγγραφα. Ο κύριος Γκέρτς όταν μετά όσα μας είπε μου θύμισε ε, μια περίπτωση που συνέρχεται ένα φίλο στα, στο μετρό φορούσε είχε τα μαλλιά, του, τα μαλλιά της, συγγνώμη, εντελώς άφρο, διάφορα χρώματα, κόκκινα, πράσινα. Και είπα, της είπα, μα τι έκανες. μου λέει, μα ε, είναι, φταίει ο, ο μου. Αυτά συμβαίνουν στο Λονδίνο και όπως καταλαβαίνετε έχουν κάποιες επιπτώσεις απρόπτες. Τώρα, ας περάσουμε στο θέμα μας πρόβαση του κοινού στα έγγραφα. Να πω ευθύς εξ αρχής πως ε, οι Σκιώδης ε, και εγώ είχαμε μια πολύ καλή και επικοδομητική συζήτηση στο Στρασβούργο όπου συζητήσαμε πολλά θέματα αλλά πρωτίστως τις αλλαγές που εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες και νομίζω ότι αυτό, αυτό συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες οι αλλαγές που είναι απαραίτητες και που θα πρέπει να εισαχθούν εν ώψη της ε, εφαρμογής της Εθνικής Λισαβόνα. Συζητήσαμε επίση ότι ο καλύτερο τρόπο για να το πράξουμε θα ήταν μέσω μιας προφορική ερώτηση. προκειμένου να γνωρίζουμε τις προθέσεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος, διότι ε, όταν λάβουμε τις πολιτικές απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή της συνθήκης, ε, μόνο τότε μπορούμε στην Επιτροπή να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα αναφορικά με τις επιλογές που θα ανοιχθούν σε εμά και οι επιλογές αυτές είναι πολλές. Πιστεύω επίσης ε, πως αυτό θα επιλύσει το ζήτημα άσχετα από την πολιτική σκοπιά του καθενός το ζήτημα της ε, πρόσβασης ε, στα έγγραφα αν αυτή θα είναι βελτιωμένη, μειωμένη και το θέμα της ε, ερμηνείας και το θέμα της διερμηνείας. η συνθήκη της Αβώνας αλλάζει το νομικό και πολιτικό πλαίσιο του κανονισμού παρέχοντας στους πολίτες μεγαλύτερες ευκαιρίε να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ένωσης. Ε, να τονίσουμε τη σημασία αυτών των αλλαγών για τις μορφωτικέ σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολίτε τη, πιστεύω πως θα ήταν καλύτερο η Κομισιόν να υποβάλει μια νέα πρόταση που θα αντανακλά της, ε, την πραγματικότητα προκύπτει μέσω τη νέα συνθήκης. αυτό θα ενισχύσει τα δικαιώματα πρόσβαση ε, των πολιτών στο Γραφείο Υπουργού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου Επιτροπή ε, Υπηρεσιών και Γραφείων, κάτι το οποίο θα βελτιώσει τη συμμετοχή των πολιτών στι δραστηριότητε. Αυτό ανέφερε ο κύριο Διαμαντούρο, ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί κομμάτι της, ε, του κανονισμού 1049 του 2001. Κυρία Πρόεδρε, Πολλά είναι τα ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αυτά, αυτές που έχουμε εδώ έχει προετοιμάσει η νομική, έχει προετοιμάσει η νομική υπηρεσία για το Κοινοβούλιο και όλοι ε, στερνιζόμαστε την παράγραφο 15 του τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα άρθρα 9, 11, 13 και 16. Θα μπορούσα να τα διατρέξω αν θέλει να διατρέξω την νομική άποψη, την, τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας, συγγνώμη, αλλά καλύτερα να αναφερθώ σε κάποιε σημαντικέ πτυχές. Η εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνας ε, θα τροποποιήσει και αυτό έχει σημασία όχι μόνο τι νομικές βάσει ε, για του κανονισμού που διέπουν την πρόσβαση στα έγγραφα αλλά και το νομικό περιεχόμενο εντός του οποίου ο κανονισμό θα λειτουργήσει ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τι σχέσει ε, ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολίτε. Αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό για το περιεχόμενο του μελλοντικού κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα. Το έβδομο εκτιμώντας αναφέρει την επιθυμία των μελών να ενισχύσουν περαιτέρω τη δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Η νομική υπηρεσία αναφέρει ότι άρθρα 11, παράγραφος 1 και παράγραφος 2 επίσης έχουν ιδιαίτερη σημασία ζητάει από, ζητούν από τα όργανα να παρέχουν στους πολίτες και στους εκπροσώπους τους να μπορούν να ανταλλάσσουν ελεύθερα ε, ε, γνώμες σε όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όλες οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι γνωστές, θα πρέπει να είναι διάφανες, διαφορετικά πώς θα μπορούν να γνωστοποιούν την θέση τους οι πολίτες. Το άρθρο 13.1 ε, ζητάει από τα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο του, ε, του των ευρωπαϊκών κανόνων να ε, φροντίσουν τα συμφέροντα των κρατών μελών και των πολιτών χωρίς να αναφέρουν το συμφέρον των θεσμικών οργάνων ως ζήτημα προτεραιότητας. Θα μπορούσα να τονίζω και άλλα στοιχεία αυτής της εξαιρετικής γνωμοδότησης, αλλά όσοι δεν την έχουν αναγνώσει, παρακαλώ και του παρατρύνω να την διαβάσουν. Θεωρώ λοιπόν από το καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε, ε, όπως είπα και στην αρχή, παρά τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις που έχουμε ή που μπορούμε να έχουμε, να διαβεβαιωθούμε ότι σε πολιτικό επίπεδο αυτά που το Συμβούλιο και η Κομισιόν προτίθεται να πράξουν να μας, καταστήσουν, να, τα καταστήσουν ξεκάθαρα. Το, η προφορική ερώτηση θα αφορά θέματα όπως ε, η αναφορά στα άρθρα που προανέφερα, επίσης ε, θα αφορούν αιτήματα σχετικά με το νομικό κενό το οποίο υπάρχει στον τομέα. Να ζητήσουμε λοιπόν από το Συμβούλιο και την Κομισιό να θεωρήσει τον κανονισμό το αργότερο πριν από το τέλος Ιουνίου 2010. Ως εκ τούτου να ζητήσουμε από τα δύο θεσμικά οργάνα να λάβουν υπόψη τους νέους κανόνες ε, της συνθήκη για την ε, διαφάνεια και την δυνατότητα αύξησης συμμετοχής των πολιτών. Αυτό που γνωρίζετε επανειλημμένα ε, στην δεύτερη τέρκο υπόθεση. Ε, εδώ σε ό,τι φορά τα εμπιστευτικά έγγραφα. Αυτά εμπίπτουν στο πλήσιο του άρθρου 4 και 9. Το άρθρο 9 αφορά τα ευαίσθητα έγγραφα. Και πράγματι υπάρχει και το, προνόμιο, το προνόμιο όπου ένα τρίτο μέρος αποφασίζει να αρνηθεί την πρόσβαση στα έγγραφα και να διατηρηθούν κάποια έγγραφα απόρριτα. Τώρα πώς αυτό το προνόμιο μπορεί να προσδιοριστεί και πώς να οριστεί προκειμένου να προστατευτούν οι πολίτες Γνωρίζω ότι τα άρθρα 4 και 9 θα ε, ε, έχουν ανάγκη από περαιτέρω αποσαφήνιση και περαιτέρω διευκρινήσεις. Χρειάζεται λοιπόν οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση για να τους διευκολύνουμε και το έργο τους. Και αυτό σε όλα τα θεσμικά όργανα, σε όλα τα όργανα μάλλον. Διότι Αυτό το σημαντικό που εισαγάγει η Λισαβόνα σε σχέση με τον κανονισμό 1049 είναι ότι δεν εφαρμόζεται πλέον στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν και στις υπηρεσίες και στα γραφεία που έχουμε δημιουργήσει εφαρμόζεται και σε ορισμένε περιπτώσεις και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Europol και στην Eurojust και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως απαιτούνται σαφείς κανόνες ειδικά με την πρόσβαση ή μη πρόσβαση σε έγγραφα. Διαφορετικά αντί να προστατεύουμε τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες τους τα αποδυναμώνουμε. Και τέλος να πω στους φίλους συνομοθέτες ότι δεν θέλω όλα αυτά να οριστούν και να προσδιορίσουν μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θέλω εμείς να τα προσδιορίσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Θέλουμε, θέλω να τα εξετάσουμε το θέμα, διότι ο κανονισμό όπως πέρασε το 2001 δεν ήταν τέλειος, άμα η νομολογία μας το απέδειξε. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω, στο ένα πνεύμα έντιμης ε, συνεργασίας ε, είναι να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ξέρουμε πως υπάρχουν προβλήματα με ζητήματα ανταγωνισμού. Ας πούμε λοιπόν στο Συμβούλιο επίσης ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα του Συμβουλίου. Που προτείνει ένα κράτος μέλος ή ένα Συμβούλιο προκειμένου να ε, ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Φροντίσουμε λοιπόν να επιλύσουμε τα προβλήματα, αλλά μην προσπαθήσετε να τα ρυθμίσετε μειώνοντας την δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα σε σχέση με τα όσα ήδη υπάρχουν στον κανονισμό 1049. Το λέω αυτό πραγματικά με στο πλαίσιο μιας έντιμης και ειλικρινούς συνεργασίας. Νομίζω ότι η συνθήκη που τα θα είναι το Μάστριχτ, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει έντιμη πολιτική συνεργασία. Αυτά τα οποία μας λεγόντουσαν εδώ και καιρό είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει κάνει ακόμα την πρώτη ανάγνωση, άρα δεν θα διαπραγματευτούμε μαζί σας. Εντυπωσιακό. Όταν ε, βλέπουμε το υψηλό ποσοστό νομοθεσίας που έχει περάσει από το σώμα μας, προτού το Κοινοβούλιο να κάνει την πρώτη ανάγνωση και μετά, από την πρώτη ανάγνωση, μετά αφού κάνει την πρώτη ανάγνωση και καταλήξει σε κάποια συνεννόηση, κάποια συμφωνία. Υπήρχε λοιπόν επιτυχία όταν ε, είχαμε μια πολύ στενή και οικοδομική συνεργασία. Ευχαριστώ για τα λόγια σας με πολύ πάθος μιλήσατε. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, πρέπει να λάβουν ακόμα κάποια βήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πραγματική κουλτούρα διαφάνειας. Νομίζω ότι και κάποια αυτοκριτική σε αυτό το νίκο, σε αυτό το σώμα επιβάλλεται. Γιατί αν θέλουμε να προβλέψουμε την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίω σε διοικητικά και οικονομικά θέματα, και εμεί οι ίδιοι, Α κάνουμε την αυτοκριτική μα, γιατί μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πολύ ωραία. Κυρία Μαρία Χέρμπε από τη Σουηδική Προεδρία θα ήθελα να σχολιάσει πολύ σύντομα όμω. Έδωσα τον απαραίτητο χρόνο στον κύριο Κάσμα, του επέτρεψα να μιλήσει παραπάνω, αλλά οι υπόλοιποι θα ήθελα παρακαλώ να σεβαστούν το χρονοδιάγραμμα. Η Σουηδική Προεδρία παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ που με επιτρέπετε να σχολιάσω το θέμα. Θα θέλαμε και εμείς ε, να συνεργαστούμε ανοιχτά και τίμια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα και νομίζω ότι το ξέρει ο κύριος Κάσμαν. Όπως είπαμε και στο παρελθόν, ε, από πλευρά Σουηδικής Προεδρίας δηλαδή, το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση πριν ε, συζητήσουμε θέματα διαφάνειας με το Κοινοβούλιο, αυτή η αναφορά δεν είναι ακριβής. Γιατί δεν είχαμε πάρει το πράσινο φως να συνεχίσουμε με βάση τα όσα είχαμε αποφασίσει το 1992. Περιμένουμε την ερώτηση που θα μας υποβάλλετε και σκοπεύουμε να απαντήσουμε σε αυτή την ε, ερώτηση. Ε, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. να είστε σίγουροι ότι είμαστε και έτοιμοι και έχουμε και διάθεση να συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί σας, μια και είναι τόσο σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη Σουηδία, η οποία πραγματικά ήταν πρωταθλητής πάντα της διαφάνειας και τώρα και στο παρελθόν και σας ευχαριστώ που ήσασταν και τόσο σύντομοι. Κομισιόν ποιος εκπροσωπείται, υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν εδώ, ο κύριος Μάς. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι τόσο σύντομο όσο και η Σουηδική Προεδρία. Ε, και η Κομισιόν είναι ανοιχτή και διατεθειμένη να συζητήσει αυτά τα θέματα. Αλλά και εγώ θέλω να επιβεβαιώσω την θέση τη Σουηδική Προεδρία. Είμαι σε μια νομοθετική διαδικασία όπου το Κοινοβούλιο δεν έχει ολοκληρώσει την πρώτη α, ανάγνωση. Ε, το Κοινοβούλιο δεν ψήφισε όμω αυτό το ψήφισμα. Είμαστε λοιπόν σε μια άτυπη συζήτηση ακόμα. Η Κομισιόν λοιπόν δεν θα λάβει σε αυτήν την ε, φάση νέα ε, πρωτοβουλία. Είμαστε μια υπηρεσιακή, θα έλεγα, κυβέρνηση μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά τη, μάλλον στι αρχέ του επόμενου χρόνου, η επόμενη Επιτροπή. Θα απαντήσει, βέβαια, η Επιτροπή στην ε, προφορική ερώτηση όποτε υποβληθεί στην Ολομέλη του Νοεμβρίου ή του Δεκεμβρίου. Και επίση, πολύ σύντομα θα κάνει τι απαραίτητε προσαρμογέ, τα απαραίτητα. Θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για το κοινοτικό και εκτιμένο. Ε, για να το ευθυγραμμίσει με τη Λισαβόνα. Ε, θα επεκτείνουμε ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογή του 1049 ε, σε όλα τα θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τροποποιήσουμε το κανονισμό και όπω είπα, νομικέ υπηρεσίε της, του Συμβουλίου αυτό είναι πολιτικό θέμα και όχι νομικό θέμα. Και επομένω, εμεί θα το προχωρήσουμε αυτό το θέμα μόνο στα πλαίσια τη επόμενη επιτροπή, τη επίσημη επιτροπή, δηλαδή. Πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντά τη λοιπόν η επίσημη επιτροπή. Έχω τρία αιτήματα για το λόγο, κυρία Σούμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν θέλω να, κάνω, να μακρηγορήσω, απλώς τα ορισμένες παρατηρήσεις γιατί ο εισηγητής έχει ε, κάνει καλή δουλειά με τις προφορικές ερωτήσεις αλλά ορισμένα θέματα πρέπει να τα αλλάξουμε διότι ο συνάδελφος Κάσμαν είπε ότι όλα αυτά δεν αναφέρονται μόνο στο άρθρο 15 της Συνθήκης Λισαβόνας αλλά και σε άλλη 12 13, 16, το 15 δεν αναφέρεται καν στο κείμενο και καλό θα ήταν να αναφερθεί. Γιατί αν διαβάσουμε το άρθρο 15 βλέπουμε ότι λέγονται πολλά για, την, ε, ε, ε, για τη Λισαβόνα. Δεν ξέρω όμως αν αυτό το άρθρο 15 μόνο του είσαι συνδυασμό με τα άλλα άρθρα επαρκεί και ίσως θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς στη διατύπωση του κειμένου αναρωτιέμαι κιόλας εάν ένα τέτοιο σοβαρός ε, κίνδυνος ενός ε, ε, δημιουργείται για, νομικό κενό ή με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ή αν είναι υπερβολική η διατύπωση αυτή και θα έπρεπε να μετριαστεί. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση διότι έχουμε συζητήσει στο Στρασβούργο το θέμα των προφορικών ερωτήσεων με τους συζητητές αλλά δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι η συνθήκη της Λισαβόλας θα ισχύσει τόσο γρήγορα μας προκατέλαβε η κατάσταση και γι' αυτό ο συγχρόνος και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπότε το ερώτημα είναι υπό αυτήν την ιδιάζουσα κατάσταση πώς θα προχωρήσουμε και καλό θα ήταν να αφήσουμε τη δυνατότητα στη νέα Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Δεν έχει πολύ νόημα μια ε, ε, απερχόμενη ε, Επιτροπή να ασχοληθεί και να επιληφθεί των θεμάτων αυτών. Υπάρχει και μία σάφια στο κείμενο της προφορικής ερωτήσεως η οποία συγχαίει την διαθεσμική διαφάνεια η οποία επιλύεται με διαθεσμικές συμφωνίες και την διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στην πληροφορία. Ίσως ε, αυτά θα έπρεπε κάπως να δουλευτούν και ε, να εκφραστούν πιο σωστά. Έχω και μία τελική ερώτηση. Στην τελευταία γραμμή ε, αναφέρεται μία οδηγία και δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η 2389 οδηγία στο κείμενο αυτό διότι 398 ε, δεν ξέρω ε, τι, ποιο είναι το νόημα διότι εδώ υπάρχουν ε, υπάρχουν διάφορα κείμενα και η οδηγία 2003, 98 του 2003 οδηγεί στο ότι συγχέουμε την κατάσταση Γι' αυτό και νομίζω ότι καλό θα ήταν να το αναδιατυπώσουμε. Αλλά είναι κάτι που πάει παραπέρα από την προφορική ερώτηση. Θα υπάρξει μία επεξεργασία και ενδεχομένως εγώ κάνω λάθος και γι' αυτό θέτω το ερώτημα του τι σημαίνει η ύπαρξη της 98 του 2003 οδηγία εδώ. Κυρία Χάουτελα, είχα μια καλή συζήτηση στο Στρασβούργο με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές και το πνεύμα ήταν ότι θα θέλαμε να θέσουμε το θέμα της πρόσβασης στην πληροφορία και στα έγγραφα ξανά, γιατί είναι ένα σημαντικό πολιτικό θέμα. Υπήρξε τεχνικό, και τεχνικό θέμα, έχει μια τεχνική διάσταση και όπως είπε και ο συγητής, ε, υπήρξαν αντιδράσεις από τα άλλα ε, θεσμικά όργανα και έγιναν και απόπειρες για να διευρυνθεί η πρόσβαση στα έγγραφα από τους πολίτες. Συμφωνούμε πάρα πολύ δηλαδή με αυτό και ελπίζουμε ότι ο κύριος Κάσμαν εξακολουθεί να είναι υπέρμαχος ενός ψηφίσματος. Γιατί χάρη σε ένα ψήφισμα μπορεί το Κοινοβούλιο να εκφραστεί για τι ε, βασικές αρχές. Γιατί το χρειαζόμαστε αυτό δηλαδή υπό την ε, Λισαβόνα. Τώρα που κοιτάζω όμως το κείμενο, μπερδεύομαι λιγάκι. Ε, συμφωνώ με την κυρία Σάμερ για αυτά που είπε. Πιστεύω ότι οι νομικές υπηρεσίες μας έδωσαν συνετέ συμβουλέ. για αυτό που είπατε ότι η προνομιακή πρόσβαση στα έγγραφα από τα θεσμικά όργανα ζητήμα χωριστό και διέπεται από διαθεσμικές συμφωνίες. Ε, έχουμε μια συμφωνία που θα αναθεωρηθεί συγκεκριμένη πολύ σύντομα από ό,τι ξέρω. Επίσης, νομίζω ότι μπορούμε να πλουστεύσουμε το ερώτημα αρκετά. Ε, και νομίζω ότι υπάρχει και ένα μπέρδεμα, μια σύγχυση στη μεσαία ερώτηση, τη δεύτερη ερώτηση για το πλαίσιο για την μεταχείριση της εμπιστευτικής πληροφορίας. Η λέξη εμπιστευτικός, εμένα με παραπέμπει τουλάχιστον, σε τέσσερις κατηγορίες διαβαθμισμένων εγγράφων, περιορισμένα, ε, εμπιστευτικά, ε, μυστικά και top secret. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήθελε ο εισηγητής να αναφερθεί σε αυτά. Ο στόχος ήταν να συζητήσουμε περισσότερο την πρόσβαση ή μη πρόσβαση. Κάτι τέτοιο, έτσι, μια, έτσι ένα γενικό διαχωρισμό. Τι σημαίνει αυτό το ιδιαίτερο προνόμιο. Ε, εγώ δεν ε, είμαι και διερμηνέας να το μεταφράσω στη γλώσσα μου, αλλά δεν έχω και την μετάφραση στα φιλανδικά για να μου το εξηγήσουν. Ο λόγος του Μάικλ Κάσμαν ουσιαστικά ε, αντανακλά αυτό που θέλαμε στην πραγματικότητα να ρωτήσουμε την Κομισιόν ε, και το Συμβούλιο. Δηλαδή την έκθεση του Διαμαντούρου και τη θαυμάσια έκθεση της νομικής υπηρεσίας. Δεν θα μπορούσαμε έτσι πολύ γρήγορα να διατυπώσουμε την ερώτηση αυτή, τη δεύτερη, τη μεσαία, ούτως ώστε να είναι τόσο τεχνική και να είναι ε, ερώτηση επί της αρχής, επί των αρχών. Απλώς να γράψουμε αυτά που μας είπε ο Μάικλ, έτσι προφορικά. Νομίζω ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να θέσουμε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Τέλος πάντων, αν κρατήσουμε αυτή τη μορφή, το πρόβλημα είναι ότι το Συμβούλιο έχει ένα πολύ εύκολο τρόπο για να παρακάμψει την ερώτηση. Θα πει, πολύ ωραία, είναι το δικαίωμα τη πρωτοβουλία. Ποιο το έχει, Κομισιόν. Α απαντήσει Κομισιόν. Τσακ, πάει το μπαλάκι. Νομίζω ότι το ερώτημα προ το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι πολύ πιο απλό, να αφορά τι βασικέ αρχέ και πολύ πιο σύντομο. το βασικό θέμα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα όμω. Ε, θα πρέπει να, να το κάνουμε και να το περίσουμε στην πιο πολιτική του διάσταση. Έτσι. Ευχαριστώ. Ε, ο κ. Ντεγιάνκ έχει το λόγο. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να σχολιάσει. Όχι, δεν υπάρχει, άρα ο κ. Ντεγιάνκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω τα είπε η κυρία Χάουταλα. Στη συνάντηση του Στρασβούργου που έγινε με τους σκιώδεις εισηγητές, η ατμόσφαιρα ήταν θαυμάσια. Και εγώ είχα πει ότι όταν μιλάμε για την πρόσβαση στην ενημέρωση για τους πολίτες, θα πρέπει να μιλάμε με καθημερινό τρόπο, με καθημερινή γλώσσα, όχι με ξύλινη γλώσσα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να επισέλθουμε σε πολύ περίπλοκες διαδικασίες και να μπερδευτούμε πάρα πολύ. Ε, και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Όταν μιλάμε για το κοινό, ε, πρέπει να μιλάμε με απλό τρόπο. Θέλω ενημέρωση, ας πούμε, για το κοινό και θα πρέπει να είναι εύκολη πρόσβαση για το κοινό και μάλιστα να έχει νόημα ε, η πληροφορία χωρίς κατά ανάγκη τον αριθμό του εγγράφου, περιττές ε, πληροφορίες. Θέλω να πάρω πληροφορίες. Και βλέπω ότι, θυμάμαι μάλλον ότι η ατμόσφαιρα στην ε, συνεδρία του Στρασβούργου ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Ε, συμπερασματικά αυτό που είχαμε πει στο Στρασβούργο ήταν ότι θα πρέπει να έχουμε σαφείς αρχές, να συμφωνήσουμε σε αυτές και όλοι να τις καταλαβαίνουν. Γιατί όταν τέτοιου τύπου φακέλους τους μεταφέρουμε, ας πούμε, ε, στην τους φανταζόμαστε μάλλον στην καθημερινότητα, θα πρέπει να φανταστούμε πώς τους καταλαβαίνει και ο απλός άνθρωπος. Συμφωνώ ε, με την ιδέα του κ. Κάσμαν, θα πρέπει να υπάρχει έτσι, πραγματική συνεργασία, τίμια συνεργασία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Το θέμα είναι πολύ επίγον. Οι εκλογές μας μας μιλάνε για αυτό το θέμα, όμως η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν το θέλουν τόσο επίγονο θέμα. Ε, συχνά μας ε, μπερδεύουν με τεχνικά επιχειρήματα, Μα λένε «Α, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση για τον α ή β περίπλοκο πάντα λόγο». Ε, θα ήθελα λοιπόν να τι αφήσουμε αυτέ τι ερωτήσει, αλλά να τις ε, διατυπώσουμε με λιγότερο ξύλινη γλώσσα. Όταν γίνει η συζήτηση δε στην Ολομέλεια, θα ήθελα να εξασφαλίσουμε ότι και τα συμπεράσματα της συζήτησης είναι πολύ κατανοητά έτσι με... και να, τα... να είναι διατυπωμένα με απλά λόγια. Πολύ ωραία. Θα δώσω ξανά το λόγο στον εισηγητή. Έγινε μια πρόταση να αναδιατυπώσουμε το προφορικό ερώτημα και να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα ε, στον τρόπο που θα απευθύνουμε το ερώτημά μας προς την Κομισιόν και στο Συμβούλιο είναι και δυνατό και επιθυμητό και καλό θα ήταν να το κάνουμε πριν την αυριανή συνάντηση το απόγευμα. Λοιπόν, μπορείτε να μας εξήγησετε όλα αυτά. Κυρία Πρόεδρε, ε, θέτετε τα ερωτήματα με τέτοιο τρόπο που <laughs> κανένας δεν μπορεί να σας πει όχι. Ε, εγώ είμαι υπέρ της συλλογική δράσης. Ε, αυτό που κάναμε το 2001 είχε ένα καλό. Συμπεριλάβαμε όλες τις νομοδοτήσεις. Ε, είχαμε μια συλλογική αντιμετώπιση. Έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Ε, εγώ είμαι έτσι καλλιτέχνη ε, και όλοι είναι όλοι οι πολιτικοί είναι καλλιτέχνε με έναν τρόπο. όταν παρουσιάζει κάτι πρέπει να έχει και το θάρρο να το να τα αλλάζει. Ε, ακούστηκαν ενδιαφέρουσε προτάσει σήμερα το απόγευμα από όλου του ομιλητέ και διαρωτώ με μήπω η Επιτροπή μου επιτρέπει να ετοιμάσω μέχρι αύριο το μεσημε... στο μεσημεριανό γεύμα την τελική διατύπωση που θα την δώσω στους σκιώδεις συζητητές εκ των προτέρων, μόλις την ετοιμάσω φυσικά, και θα διαγράψω οποιαδήποτε περίπλοκη ορολογία, αλλά όμως θα συμπεριλάβω και όλα τα καθόδη θέματα. Δηλαδή, της υγείας σας θα πρέπει να είμαστε και ορθολογικοί, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ξεχνάμε και ποια είναι η νομική βάση. Ε, θα πρέπει να αναφέρω δηλαδή τα συναφή άρθρα. Ε, επίσης, ε, έχετε δίκιο που είπατε ότι ήταν μεγάλη παράληψη το άρθρο 15, που το ξέχασα να το πω. Τώρα, τι να σας πω, Σουηδική Προεδρία. Ε, θα σας πω κάτι και το νο. Εγώ έχω συνεργαστεί με τη Σουηδική Προεδρία το 2000-2001 για να υλοποιηθεί εκείνο το μέτρο. Ξέρω τι δουλειά κάνετε, τι δυσκολίες έχετε ως Προεδρία. Τώρα είσαστε στην Προεδρία του Συμβουλίου. Το λέω αυτό στο Μάρκ. Και στην Κομισιόν δηλαδή. Ε, δεν είναι... Δεν μας αρκεί να μας λέτε. Είσαστε νέο κοινοβούλιο. Δεν έχετε τελειώσει την πρώτη σας ανάγνωση. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Γιατί μέχρι την ψηφοφορία που κάναμε το Μάρτιο ε, και, τότε τα ίδια μας λέγατε. Και μετά, και μετά μας ξαναείπατε τα ίδια. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε μαζί σας. Ε, η νομική υπηρεσία μας λέει δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε μαζί σας γιατί το κοινοβούλιο δεν έχει θέση. Αυτό το λένε οι άνθρωποι που είναι απρόθυμοι και συντηρητικοί προς τις αλλαγές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε αυτό το θέμα. Να... Για όλους μας, για όλους τους εμπλεκόμενους. Άκουσα τι είπατε, το σημείωσα, αλλά δεν είναι απόλυτα αληθές. Η ίδια δικαιολογία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Καλή η δικαιολογία, αλλά πρέπει να ξεπεράσει τι δικαιολογίε αν θέλετε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ όλου όσου ε, συμμετείχαν. Ε, θα προσπαθήσω να το χτενίσω το κείμενο και σας υπόσχομαι να επανέλθω μέχρι τις 11. Το λέω έτσι, είναι μια προκαταρτική ώρα, έτσι. Και θα καθορίσουμε και μια προθεσμία μέχρι τις 12.30. Εντάξει, όλα αλλάζουν, έτσι. Αλλά θα προσπαθήσουμε να ε, συμφωνήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Όπως είπε και η Χάιντι εξάλλου, ξέρω πολύ καλά ότι αυτό που μετράει είναι το πώς επιλύουμε αυτό το θέμα χωρίς ψήφισμα. Um, Ευχαριστώ πολύ. Υποθέτω πως γίνεται δεκτή η πρόταση του εισηγητή σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Θα φροντίσουμε όλοι λοιπόν να τον βοηθήσουμε και να υποβάλουμε γραπτός κάποια σχόλια ευθύς αμέσως ενδεχομένως μετά το πέρας της η νομική υπηρεσία είπε στο Συμβούλιο, όπως είπε η ότι δεν υπάρχει βάση προς για διαπραγμάτευση. Όπως και στο θέμα... όπως και στο θέμα της, του SWIFT με τους Αμερικανούς θερμονομικής βάσης. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο της μεσαίας διατάξεως. Μάικλ. προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ε, νομική βάση αυτό που είπα στην αρχή. Επειδή δεν θυμάμαι πλέον τι είπα, διότι ξέρω ότι κανείς μιλάει με αυτά, σύμφωνα με αυτά που αισθάνεται, θα ζητήσω λοιπόν να δοθεί μια ταινία μαγνητοφωνημένη για τα όσα είπα σήμερα το απόγευμα. Εντάξει, ελπίζουμε να δείξει το ίδιο πάθος ε, και αύριο και όλα θα γίνουν απόλυτα κατανοητά Τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο της μισής διατάξεως και ίσως θα μπορούσαμε να το ολοκληρώσουμε σύντομα διότι επανειλημμένα το, μάλλον το συζητήσαμε πριν μερικές εβδομάδες το δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης σε ποινικέ διαδικασίες. Ε, πρόκειται για μια πρόταση που αφορά τα τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι του όλου πακέτου επί του οποίου έχει ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να σας πενθυμίσω που τού να δώσω το λόγο στην συγκεντριά μας την Βαρόνη Σάρα που πρόκειται για μια πρόταση που άπτεται του τρίτου πυλώνα και θα επηρεαστεί άμεσα με την θέση ισχύτηση της Συνθήκης Λισαβόνας και Τώρα φτάνουμε στη ζήτηση που είχαμε στις αρχές του απογεύματος. Σάρα, σου δίνω το λόγο ζητώντα σου παράλληλα να είσαι λακωνική προκειμένου να το ολοκληρώσουμε σύντομα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ε, δεν θα χρειαστεί στον να πω ότι άλλες ε, εκθέσεις όπου οι παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους. Ε, ναι, πριν από μερικές εβδομάδες υπήρχε μια πρώτη ανταλλαγή απόψε. Εγώ τώρα έχω συντάξει την τελική μου έκθεση και ίσως να πρέπει να εξηγήσω κάποια από τα βασικά σημεία της εκθέσεως. Ίσως να μου χρειαστεί ένα λεπτό να το πράξω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σε αυτήν την ενδιαφέρουσα φάση όπου θα τεθεί σε ισχυρή 1η Δεκεμβρίου η Συνθήκη Λισαβόνα. Προτού να επανέλθω στο το θέμα, να υπενθυμίσω πω ε, είναι σημαντική αναβάθμιση των ε, δικαιωμάτων ε, κάτι το οποίο επανειλημμένα τόνισε το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια. Όπως ε, γνωρίζετε, εδώ υπήρξε μια προσέγγιση βήμα προς βήμα και το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει σε πολιτικό επίπεδο για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα τον οδικό χάρτη, ο οποίος λέει ότι θα τα ολοκληρώσουμε αυτά τα ζητήματα το ένα μετά το άλλο, αυτή είναι η πρόθεσή μας και το δεύτερο είναι η οδηγία πλαίσιο για τη διερμηνία και τη μετάφραση. Και το τρίτο είναι ένα ψήφισμα για τι πρακτικέ επιπτώσει εφαρμογή αυτή τη οδηγία, τη απόφαση, και είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο που δεν ζητήθηκε η γνώμη μα για τα υπόλοιπα δύο θέματα. Χρειάζονται λοιπόν αυτά τα δικαιώματα διερμηνία και μετάβραση, αλλά χρειάζεται επίση και η νομική αρρωγή κλπ. Θα σας αναφέρω κάτι τώρα, μια περίπτωση ενό ε, ε, πολίτη της εκλογική περιφέρειας, ο οποίο πάει στην ε, Ελλάδα επέστρεψε και ασκήθηκε έφεση το Σεπτέμβριο και ο κατηγορούμενος ένα μήνα αργότερα ε, του έμαθε ότι του αρνήθηκαν την ε, αποφυλάκηση μέσω εγγύησεως και αυτή η απόφαση είχε γραφτεί στα ελληνικά. Μολονότι είχαν διεύθυνση ε, κατοικίας στην Ελλάδα διότι είχε συγγενείς που ζουν στην χώρα αυτή. Με συμπτώσει δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά με συμπτώσει και η μετάφραση. Μα η κατάσταση τα ζητήματα μετάφραση δεν είναι διόλου ικανοποιητική. Και επίση υπάρχει και το θέμα του ε, Ευρωπαϊκού Εδάλματο Σύλληψης, το οποίο εμπλέκεται στην περίπτωση αυτή της ε, μετάφρασης. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η προσέγγιση βήμα προς βήμα και θεωρήθηκε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να προχωρήσουμε. Η έκθεσή μου αναφέρεται σε, κάποιες, ε, σε κάποια ζητήματα που μόλις ότι η πρόταση Κομισιόν είναι καλή, μεν θα μπορούσε όμως ε, να βελτιωθεί, να ενισχυθεί περαιτέρω όπως η επέκταση του δικαιώματο ε, να καλύπτονται όλα τα στάδια της ποινική διαδικασίας συμπεριλαμβανομένως και της ε, διαδικασίας που ακολουθεί την ε, σύλληψη, την κράτηση, η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία, δεν έχει εκδικαστεί υπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν οι αρχές να ενημερώνουν τους υπόπτου και θα πρέπει να ενημερώνονται φυσικά γραπτός ο κατηγορούμενος. Χρειάζεται λοιπόν να αναφέρουμε εδώ την ε, ανάγκη στο δικαίωμα της διερμηνίας και της μετάφρασης ε, στις ποινικέ αυτέ διαδικασίες. Και Και κάτι ακόμα τώρα. Το ζήτημα της άρνησης παροχής διερμηνίας και μετάφρασης ε, θα πρέπει να αιτιολογείται διόντως. Και τέλος, τονίζω πως θα πρέπει να υπάρχει και ένας κατάλογος ανεξαρτήτων διερμηνέων και μεταφραστών διαθέσιμων στα δικαστήρια. Προσπάθησα λοιπόν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πάντως, δεν ξέρω αν θα μπορέσει το Συμβούλιο να υιοθετήσει αυτά τα μέτρα πριν από την 30 Νοεμβρίου. Για μα η περίοδο ε, τρίμηνη ολοκληρώνεται πριν από τι διακοπέ των Χριστουγέννων και το χρονοδιάγραμμά μας αναφέρει ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί την συνολομέλεια του στην και να και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμά μας διότι δεν προβλέπεται κάποια συνεδρία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ πέραν των διαφόρων ακροάσεων που έχουν προβλεφθεί. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτό θα εμπέσει στον κατάλογο των μέτρων που η Κομισιόν θα υποβάλει στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και ελπίζω πως δεν θα χάσουμε τον ρυθμό μας, την τάση που έχουμε αποκτήσει και ελπίζω η Κομισιόν να μπορέσει να συμπεριλάβει σε εργασίες της ε, την ε, δουλειά που έχουμε κάνει. Είχα συνάντηση με τον σκιώδη Σιγητή χθε. Και πιστεύω δεν πρέπει να χάσουμε περαιτέρω χρόνο λόγω των νέων διαδικασιών που προβλέπονται στη Λισαβόνα και η Επιτροπή εξετάσει κατά πόσο θα πρέπει να εκφέρουμε γνώμη με τη θέση ισχύ της Λισαβόνας επί του συνόλου του ζητήματος ε, εχομένως ε, να καταθέσουμε ερωτήσεις προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα. Περιμένουμε φυσικά την ε, νέα, τη σύσταση της νέας Κομισιόν Μπες περιπτώσει ο Επίτροπος Αρμόδιος για Δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έχει πολλά να κάνει για το ζήτημα αυτό. Το Συμβούλιο έχει φτάσει σε κάποια συμφωνία η οποία μπορεί να μην είναι τόσο προοδευτική όπως θα επιθυμούσαμε. Η Κομισιόν θα μπορούσε να προωθήσει την πρότασή της η οποία πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη από την αρχική και να πείσουμε το Συμβούλιο να δείξει κάποια ευελιξία σχετικά με τα μέσα τα όσα μπορούσε να συμφωνήσει ή ακόμα και να προχωρήσει σε μια προσέγγιση βήμα προς βήμα, αν και δεν θα ήθελα να κλείσω με αυτήν την άποψη. Δεν βρισκόμαστε, βρισκόμαστε μάλλον στο πλαίσιο μιας αβεβαιότητας ε, και το σίγουρο είναι ότι το πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί υπό τον τρίτο πυλώνα αλλά είμαι αισιόδοξη και ελπίζω να υιοθετήσουμε ένα πολύ καλό μέσον. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ομιλητές στον κατάλογό μου, αλλά καταρχήν θα έλεγα τέσσερις ομιλητές. Να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά το Συμβούλιο με αυτή τη σειρά και μετά να ανοίξει η συζήτηση. Έχουμε την κυρία Κάρονα Μόργκεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι η πρώτη που θα παρέμβει. Θα ήθελα απλώς να πω ότι πολύ ε, εξετίμησα την εργασία της Βαρόνης Λάτφορντ στο θέμα αυτό. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ καιρό να συμφωνήσουμε και στις 31 Οκτωβρίου όταν καταφέραμε ε, να βρούμε μία συμφωνία ισοσκελισμένη με προστιθέμενη αξία ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι διότι έτσι υπάρχει ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ καλό. Ήταν ένας φάκελος πολύ δύσκολος, αλλά όσον αφορά το μέλλον δεν ξέρουμε πώς τα πράγματα θα προχωρήσουν με την μετάφραση και την διερμηνία αλλά υπάρχουν τέσσερα νομοθετικά μέτρα τα οποία έχουν ουσιαστικά συμφωνηθεί και ε, θα συνεργαστούμε ε, με ε, το Κοινοβούλιο για τον καθορισμό των μελλοντικών μέτρων. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω το Συμβούλιο την κυρία Βέμπερ. Το, το μικρό μου όνομα είναι πολύ δύσκολο να το προφέρετε γιατί δεν είναι σουηδέζικο. Αυτό είναι που είπα και εγώ προηγουμένως στη συζήτηση της Λισαβόνας. Είναι ένας από τους φακέλους που δεν προτείνουμε να υιοθετηθεί με το παρόν καθεστώς και προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Συμβούλιο επί του θέματος αυτού ε, η Επιτροπή θα το προωθεί αλλά όταν το Κοινοβούλιο θα υποβάλει την πρόταση με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να την προωθήσει στο Συμβούλιο και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον το, το Κοινοβούλιο θα πρέπει με τον, άλλο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε υπό μορφή ψηφίσματος, είτε υπό άλλη, να το υποβάλει στην Επιτροπή προς έλεγχο της πρότασης. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και καλή συνεργασία και ε, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε διότι αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουμε δηλαδή βαθμία να απομονώσουμε τα άλλα θέματα τα οποία μπορεί να αποδυναμώσουν ένα κείμενο ε, εάν παραμείνει στο σύνολό του θα είναι όντως ένας εξαιρετικός τρόπος να έχουμε προστιθέμενη αξία και ελπίζουμε ότι έτσι θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θέλουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μία ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώματα το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε γρήγορα ε, από τις διάφορες φάσεις για να υιοθετηθούν όλα τα θέματα όσο δυνατόν πιο γρήγορα ακόμη και αν ισχύσουν με το καθεστώς της νέας συνθήκης. Προσβλέπουμε λοιπόν στη συνεργασία που θα έχουμε μαζί σας στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Έχω στην, στο κατάλογο μου την κυρία Ρομέρο Λόπες πρώτα. Ευχαριστώ, ναι, πράγματι. Θεωρούμε πως θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δεδομένου το ότι σημείο αυτό θα περάσει σύμφωνα με τη διαδικασία της ε, Λισαβόνας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια κοινή πρόεδρος ψηφίσματος. Ε. Αρχικά είχε υπάρξει σχεδόν ομοφωνία θα έλεγα στο πλαίσιο των πολιτικών ομάδων ε, προκειμένου να προωθηθεί αυτό το δικαίωμα στην διερμηνία και μετάφραση στο πλαίσιο του οδικού χάρτη ενό ε, πακέτου που αφορά στις ποινικέ διαδικασίε και που αποτελεί το σύνολο των ε, εγγυήσεων που θα πρέπει να προωθήσουμε και να εφαρμόσουμε σε μια Ευρώπη της δικαιοσύνης και όχι μόνο Ευρώπη της ασφάλειας. Για τον λόγο λοιπόν αυτό το ψήφισμα είναι σημαντικό και θα μπορέσει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την νέα Επιτροπή, για τον νέο αρμόδιο επίτροπο που θα αναλάβει το θέμα αυτό. Θα πρέπει να θεωρήσει ότι η συμφωνία στο Κοινοβούλιο αποτελεί την βάση προκειμένου να υποβάλει μια νέα πρόταση, διότι το ζήτημα είναι πως ε, το σκηνικό έχει αλλάξει. Το σκηνικό τώρα δεν είναι πλέον το ίδιο που υπήρχε όταν ξεκίνησε η όλη συζήτηση αυτή, η οποία ξεκίνησε προκαιρού, αλλά δεν είναι και το αυτό σκηνικό όταν ε, τα πράγματα με τη Σουδική Προεδρία προχώρησαν. Η πολιτική κατάσταση λοιπόν μπορεί να κάνει να θεωρεί κανείς ότι πρόταση μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Το να επιτευχθεί φυσικά η ομοφωνία από τα κράτη-μέλη είναι κάτι το δύσκολο. Αλλά το κείμενο της 23ης Οκτωβρίου είναι ένα κείμενο το οποίο εισαγάγει και κάποιες ε, άλλες πτυχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, ε, από τη νέα πρόταση. Δηλαδή να προσπαθήσουμε ότι κάποιες θέσεις που αποτελούν οπισθοδρόμηση να εξεταστούν από μια άλλη οπτική γωνία, δεδομένου ότι το σκηνικό, όπως προείπα, είναι καινούριο, είναι διαφορετικό. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα δείχνει ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου και αυτή να ληφθεί υπόψη από την Κομισιόν και να εισαγάγει αυτό το δικαίωμα στη μετάβαση και διερμηνία ως ε, τμήμα του ολικού, της συνολικής δέσμης, του ολικού πακέτου. Το πιο λογικό λοιπόν θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει ευελιξία και ταχύτητα σε κάθε μία από τις φάσεις. Το πιο εύλογο θα ήταν να έχουμε μία οδηγία για, όλα τα, για όλη την ποινική διαδικασία αλλά υπήρξαν όπως ξέρουμε δυσκολίες ε, που ήταν προφανείς. Στο Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την άποψη ότι αυτά τα ε, δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν ένα πακέτο, μία δέσμη και οι οδηγίες μπορεί να μην είναι ενωμένες να αποτελέσουν μία, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε με τον οδικό χάρτη της Ουδικής Προεδρίας και οι οδηγίες αυτές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποτελέσουν τον δέσμη για τα δικαιώματα στην ποινική διαδικασία έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση για την οποία η συνάλφος Λούτφορτ, η συγκήτρια, που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά να μπορέσει να συνδυαστεί αυτή με την ε, νομική αρρωγή, την ε, επικοινωνία με τις οικογένειες, με τις ε, προξενικές αρχές κλπ. Θεωρούμε λοιπόν πως εάν η Κομισιόν ακολουθήσει τις υποδείξεις του ψηφίσματος θα μπορέσει να υποβάλει πρόεδρε στο Συμβούλιο, η οποία θα αποτελέσει την βάση για μια Ευρώπη της δικαιοσύνης και όχι μόνο της ασφάλειας. Ευχαριστώ κυρία Αντωνέσου, που έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω την κυρία Σάρα Λάντφορτ για τη διάθεσή της να συνεργαστεί σε αυτή τη Λυπάμαι που η έκθεση δεν ακολούθησε την συνήθη διαδικασία. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Αυτή η πρόταση είναι πλήρης. Οι τροπολογίες αφορούν τα ουσιώδη σημεία της πρότασης. Η έκθεση αυτή αφορά τα πιο σημαντικά, όπως είπα, σημεία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια από τα πιο σημαντικά σημεία και που υπάρχουν στο σχέδιο της έκθεσης. Θα τα αναφέρω αφορά την τροπολογία καταρχήν, ένα από τα σημαντικά σημεία είναι η τροπολογία 1, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να μειώσουν τα πρότυπα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα, οι τροπολογίες 4, 4 και 16 είναι πολύ σημαντικές. Πρόκειται για άτομα με ειδικέ ε, ανάγκες και μειωμένε ε, πνευματικές ανάγκες, θα πρέπει οπωσδήποτε να τα υποβοηθούμε αυτά τα άτομα. Οι τροπολογίες προσδιορίζουν το είδος της αρρωγής που πρέπει να τους προσφέρουμε. Η τροπολογία 8 που συμπληρώνει πολύ σημαντικά το δικαίωμα της ε, διερμηνίας σε όλες τις φάσεις της ποινική διαδικασίας. Μια και η κυρία Λάτφορντ υπογράμισε πολλά προβλήματα που υπάρχουν στις δικές μου τροπολογίες εστιάζω τελικά ε, σε στοιχεία που αφορούν την ποιότητα της μετάφρασης και της διερμηνίας. Αυτά ούτως ή άλλως αναφερόταν και λεπτομερώς στο ψήφισμα του Συμβουλίου που συνοδεύει την πρόταση των κρατών μελών. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να αναφέρονται και στην πρόταση απόφασης. Γιατί το να εξασφαλίσουμε ποιοτική διερμηνία και μετάφραση είναι εκ των όνου κάνευ σε όλε τι ε, φάσει τη διαδικασία. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εισαγάγουν ένα μηχανισμό ελέγχου της διερμηνία και της μετάφραση, καθώ και ένα σύστημα επιστοποίηση ε, των διερμηνέων και μεταφραστών ε, στις ποινικέ δίκες. Σε επίπεδο τώρα κράτους μέλους θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα επαγγελματική κατάρτιση, συνεχού κατάρτιση για τέτοια θέματα. Όπως είπαμε και στη σημερινή συνεδρίαση, ε, η κατάσταση είναι αρκετά ιδιάζουσα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας για την απάντηση που μας έδωσε, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω εξηγήσεις. Και θα θέλαμε να τις έχουμε γραπτός μάλιστα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας ε, και μέσα σε καλές συνθήκες μέχρι να τεθεί ε, σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Προηγουμένως από την παρουσίαση του Συμβουλίου κατάλαβα ότι αυτά τα δικονομικά δικαιώματα, για αυτά τα δικονομικά δικαιώματα δεν θα αποφασίσουμε μέχρι τις 30, τις 30 Νοεμβρίου. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει νέες προτάσεις, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια χρονική στιγμή. Και, και επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα ήθελα να γίνει τους επόμενους μήνες ε, να κάνει την πρότασή τη δηλαδή η Κομισιόν. Επίσης θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε και ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη ε, διαδικασία να την γενικεύσουμε. Δηλαδή τότε το Κοινοβούλιο <laughs> στο τέλος του χρόνου τελικά ε, αποκρισταλώνει ε, όλη τη δουλειά που κάνει σε μία σειρά από προφορικές ερωτήσεις ε, προς το, Κοινοβούλιο και, προς το Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν. Νομίζω ότι καλύτερα τα ψηφίσματα. Από σεβασμό προς την κυρία Λάτφορντ πιστεύω ότι όταν η Κομισιόν θα κάνει την πρότασή της θα λάβει υπόψη και την πρόταση του Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα τις δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ. Εάν ε, με κατηγορούσαν ε, στο δικαστήριο για ένα έγκλημα θα ήθελα να μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου άρα και εδώ δεν θα έπρεπε να <clears throat> χρειαστεί να μιλήσω αγγλικά. Ε, βλέπω όμως και δεν υπάρχει γλώσσα οπότε συνεχίζω αγγλικά. Υπάρχουν φιλανδικά? Όχι. Οπότε μην χάνουμε χρόνο. Συμφωνούμε με την άποψη της Άρα Λάτφορτ. Πιστεύουμε ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι ε, μία βαθμιαία προσέγγιση είναι καλύτερη και ότι όταν το Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα συναπόφαση θα είμαστε στο σωστό δρόμο και επιπλέον ε, όντως χρειάστηκε να ε, ε, υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη στα δικαστικά μας συστήματα. Υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη αλλά όχι η ιδέουσα βάση. Άρα χρειάζονται τουλάχιστον ελάχιστοι κανόνες και χαιρετίζουμε τις τροπολογίες. Θα θέλαμε επίσης να πούμε ότι το κείμενο αυτό εάν υιοθετηθεί θα αποτελέσει μια καλή πρόταση για τη βάση για την Επιτροπή να προβεί σε μια βελτιωμένη πρόταση και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο ε, θα επιταχύνει τη διαδικασία της εφαρμογής των διαδικαστικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ την κυρία Λότφορντ για τις εργασίες της και ελπίζω πως όλα αυτά θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο νέων διαδικασιών που προβλέπει η Λισαβόνα. Θα ήθελα να τονίσω την σημασία αυτής της ε, νομικής βάσης που θέτει η Σάρα Λότφορντ για να δικαιολογήσει τα μέτρα η βάση αυτή διαφέρει σε σχέση με την βάση της αρχικής πρότασης που έχει υποβάλει η Κομισιόν. Τώρα, ε, και επαφιόταν στην βούληση των κρατών μιλών και στην ε, εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να αποδίδουν στις διαδικασίες. Πάντως η πρόταση της ε, Βαρόνης Λάτφορντ μιλάει για τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και τα άλλα δικαιώματα διερμηνίας και μετάβασης σε ποινικές διαδικασίες. Τώρα βασιζόμενοι στην θλιβερή εμπειρία που έχουμε στη χώρα μας αλλά που υπάρχει και σε άλλα κράτη-μέλη είναι απαραίτητο λοιπόν αυτά τα μέτρα να προκύψουν από αποφάσεις ε, που θα έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι διαφορετικά οι δικαστικές εθνικές αρχές θα έχουν μεγάλες δυσκολίες στο να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση που είναι ζωτική σημασίας για να εγγυηθούμε δίκες, δίκες. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία κρίνω όπως ε, έχει το ότι πρέπει να κοινοποιούνται τα δικαιώματα στους ε, κατηγορούμενους αλλά επίσης ε, και θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος για τις ακροάσεις τις οποίες έχει στον η διερμηνία και η σημασία παράλληλα Ενό καταλόγου με εξειδικευμένου διερμηνείς τώρα. Ε, τώρα, σε ό,τι φορά 26, αυτή προβλέπει κάτι παρόμοιο, ότι αναφέρεται σε ένα εθνικό κατάλογο με εγκεκριμένους πιστοποιημένους μεταφραστές και διερμηνείς και δεν ξέρω το κατά πόσον ε, θα πρέπει να αναφερθούμε σε διασυνοριακό επίπεδο. Αλλά καλό είναι να υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός κατάλογος, ένα ευρωπαϊκό μητρό. Διότι συχνά μπορεί να προσφεύγουμε σε άλλο κράτος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ε, κατηγορούμενο, κύριο Σταβάρη. Ο τελευταίος... Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Παρακολούθησα τις τελευταίες συνεδριάσεις που διοργάνωσε η Σάρα Λάτφορντ και μου δημιουργήθηκε έτσι η γενική εντύπωση ότι ε, υπήρχαν τρεις βασικές αρχές που δεν πρέπει να λησμονούμε σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν μάλλον τρεις βασικές αρχές. Ότι ένας πολίτος, πολίτης και ύποπτος θα πρέπει να είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας. Αυτό είναι το αντικείμενό μας. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει α, πότε χρειάζεται ε, μετάφραση και διερμηνία. Αν υπάρχει κάποιος αυτό είναι ο ενδιαφερόμενος, ο ύποπτος. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το πει για αυτόν. Δεύτερον, οι διαδικασίες. Ε, όπως είχαμε πει και προηγουμένως στην προηγούμενη συζήτηση ε, για την πρόσβαση των δεδομένων, αυτό που είναι σημαντικό είναι η διαφάνεια. Αν υπάρχει διαφάνεια, όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Επομένως, και εδώ, η σωστή ενημέρωση για την ποινική διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνία αν εμπλέκονται σε ποινική δίκη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις νομές Πολιτείες, συγγνώμη, Φερρυπίν, υπάρχουν τα δικαιώματα Μιράντα. Και ο κόσμος γνωρίζει τα δικαιώματά του. Υποστηρίζω λοιπόν την κατεύθυνση προς την οποία οδηγούμαστε. Αυτό είναι το βασικό. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Πολύ ωραία, τον παλάκι ξανά στην εισηγήτρια. Σας ακούμε. Ευχαριστώ ευχαριστώ για όλους όσους συμμετείχαν. Εκτίμησα όλα τα σχόλια και την υποστήριξη από τους συναδέλφους και νομίζω ότι ακούσαμε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι δεσμεύονται και εκείνοι να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό για αυτό το φάκελο. Προφανώς εκτιμώ το γεγονός ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση στο Συμβούλιο ε, το να βρεθεί ομοφωνία. Στο μέλλον όμω δεν θα χρειαζόμαστε ομοφωνία, επομένω αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα δεδομένα. Επίσης, ε, προηγουμένως είπα ότι ίσως να υπάρχει περιθώριο ευελιξίας. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τους οποίους συναντήθηκα στο Στρασβούργο. Ε, θα καταλάβετε από διάφορες τροπολογίες μου πόσο με ενδιαφέρει να εξασφαλίσω ότι δεν υποσκάπτουμε τη σύμβαση του Στρασβούργου και την ομολογία του Στρασβούργου. Βασιζόμαστε σε αυτήν και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε τη δουλειά που έχουν κάνει στο δικαστήριο του Στρασβούργου στα πλαίσια της σύμβασης. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το σεβασμό της σύμβασης. Ε, λοιπόν, ήταν στη διάθεσή μου στι συναντήσει υπάλληλοι του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Συνολικά, λοιπόν, καλό θα ήταν να ψηφίσει η Επιτροπή για να υιοθετήσουμε την έκθεση, αλλά δεν νομίζω ότι και νομικά είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Ε, η πρώτη μα συνεδρίαση θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου. Η επόμενη δηλαδή. Και όχι απλώς δεν θα, δεν θα υπάρχει νομική ισχύ, αλλά δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε έκθεση στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα δεν θα υπάρχει πλέον τρίτος πυλώνας από 1η Δεκεμβρίου. Επομένως, μοιραία η έκθεσή μου δεν θα ε, ψηφιστεί τότε. Αλλά ίσως ε, δεν θα ψηφιστεί. Ε, ίσως όμως κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που έχουν διαβάσει την εκθέσή μου να έρθουν ας πούμε, και να μου πούνε «Α, ξέρεις, αυτό το σημείο θα μπορούσε να το βελτιώσεις». Ε, επομένως, θα έχουμε το χρόνο να τα ξαναδούμε. Αλλά ελπίζω ο χρόνος να μην είναι ατέρμονος. Ελπίζω να είμαι και η συγγήτρια στην ε, επόμενη έκθεση, η οποία θα είναι έκθεση Ladford Report 2. Κοιτάξτε, εγώ για τα οργανωτικά είμαι τραγική. Δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει πιο πολύ πολιτική. Αλλά δεν θα διερωτώ Μια και δεν μπορούμε νομικώς πώς να υιοθετήσουμε μια θέση, δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι μια κατευθυντήρια γραμμή στην Κομισιόν, ας πούμε. Ε, μέσω ενός ψηφίσματος, Φερρυπίν. Ναι. Ίσως μίλησα πολύ γρήγορα. Θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε μια τέτοια άγουσα. Αλλά καλό θα ήταν να το αφήσουμε πρώτα στους συντονιστές να το συζητήσουν. Θα ξεκαθαρίσει κάπως η εικόνα και θα ξαναδούμε το φάκελο αυτό μετά το πέρα συνεδρίες των συντονιστών και τι συμβουλή θα μας δώσουν. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, ένα ψήφισμα ενδεχομένω ε, ή με ένα προφορικό ερώτημα στην Ολομέλεια προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Ίσως καλύτερα ψήφισμα. Με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να μεταλαμπαδεύσουμε το περιεχόμενο των ιδεών του Κοινοβουλίου που υπήρχε στην εκθεσή μου. Ευχαριστώ γι' αυτό. Άκουσα όλες τις συνεισφορές. Ε,